Καλημέρα σας. Ξεκινούμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Πρώτα απ' όλα, όπως όλοι γνωρίζετε, ο τέταρτος αντιπρόεδρος, ο κύριος Χάρπορ, έχει οριστεί υπουργός άμυνας της Φιλανδίας. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι το Σεκρετό του παρετήθηκε των καθηκόντων του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κύριο Νίλ Τόρβαλτ τον αντικαθιστά. Θερμό όρισμα, λοιπόν στην Επιτροπή Αλία προ τον συνάδελφο. Κανονικά πρέπει να θέσουμε σε ψηφοφορία βέβαια την ε, αντικατάσταση του κύριου Χάγκλουντ από τον ε, κύριο Τόρβαλτ και θα το κάνουμε μετά το σημείο 4, αφού δηλαδή εγκρίνουμε την μέτρια διάταξη. Σε σχέση με τη Μέσια Διάταξη θα κάνουμε κάτι το οποίο αρχίζει να γίνεται συνήθεια και καλό θα ήταν να πάψει να γίνεται συνήθεια. Κάθε φορά αφού έχουμε καταρτήσει τη Μέσια Διάταξη αρχίζουν να έρχονται τηλεφωνήματα, επιστολές που ζητούν αλλαγή στα σημεία της Μέσης Διάταξης, διάφορες αλλαγές. Κανονικά ε, δέχομαι Συνήθως δέχομαι τα αιτήματα αυτά για τροποποίηση. Απλά έχει ξεπεράσει κάποια όρια ε, αυτή η κατάσταση και διαταράσει και τις εργασίες της Επιτροπής μας. Δηλαδή, δεν μπορεί κανείς να παρακολουθεί στη μέση διάταξη εφόσον την αλλάζουμε συνέχεια. Αυτό που λέω απλά είναι ότι αν κάποιος αλλά αν είναι απολύτως απαραίτητο μόνο νιώθει την ανάγκη, έχει ανάγκη να προτείνει αλλαγή της μέσης διάταξης, σας παρακαλώ να το πράττει πολύ νωρίτερα, να μας ενημερώνει άμεσα, διότι δεν πρόκειται να δεχθώ καμία άλλη αλλαγή της μερίσια διάταξη εάν δεν γίνει αυτό πολύ πριν από την συνεδρίαση. Και πρέπει να σας πω ότι και πάλι δύσκολο αυτό δεχτώ γιατί δεν μπορούμε να τροποποιούμε τη μεσιά διάταξη. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο, ενώ αντίθετα πριν γίνει η συνεδρία ξέρουμε ποια είναι τα ημερομηνία των συνεδριάσεων. Βέβαια, αυτοί που το κάνουν αυτό ίσως δεν είναι παρόντες σήμερα, ε, αλλά τέλος πάντων, ε, εγώ θέλω να σας πω ότι ξέρετε ε, εγκαίρως πότε είναι οι συνεδριάσεις μας και σας παρακαλώ να σέβεστε την Επιτροπή Αλίας όλοι, διότι τελικά φαίνεται σαν να μην της δίνουμε αξία. Και πάντα να υπάρχει κάτι πιο σημαντικό. Γιατί πολλοί δεν έρχονται καν στις συνδρέες Αλίας. Είναι κακό αυτό για όλους. Έχουμε και κάποιες τώρα τροποποίησεις, όπως έλεγα στην ημερήσια διάταξη, το σημείο 17 Φερέιρα και το 18, το θα τα συζητήσουμε σήμερα. Αντί των σημείων 9, την έκθεση της κυρίας Πατράου δηλαδή, του σημείου ναι, που θα συζητηθεί αύριο μετά το 19. Θα μπει μεταξύ 19 και 20, άρα 17 και 18 σήμερα και 9 αύριο, μεταξύ του 19 και του 20. Αν συμφωνείτε μπορούμε να εγκρίνουμε αυτή την αλλαγή και εγκρίνουμε και την ίδια διάταξη. Σημείο 2. Έγκριση των πρακτικών τη συνεδρίασης τη 30η και 31η Μαου. Όσοι ήθιστε θα θεωρηθεί ότι εγκρίνεται αν δεν υποβάλλει ή προβάλλει κανεί ένσταση στη διάρκεια τη συνεδρίασή μα. Ανακοινώσει του Προέδρου. Με βάση τον κανονισμό και επαληθεύσαμε ότι υπάρχει μία πρόταση από την πολιτική ομάδα Άλντε που προτείνω σαν τέταρτο αντιπρόεδρο τον κύριο Νίλς Τόρβαλς. Υπάρχει άλλη πρόταση. Εσείς ο ενδιαφερόμενος δέχεστε. Ωραία. Άρα αν δεν υπάρχει αντίρρηση, πληρούνται προϋποθέσεις ε, και διαβοής εγκρίνεται. Ορίζεται τέταρτος αντιπρόσωπος ο κύριος Τόρβαλς. Και παρακαλώ, ελάτε να καθίσετε στο Προεδρείο. Επίσης, θα ήθελα να σας ανακοινώσω καλή τύχη, κύριε Τόρβαλς, ότι η κυρία Ισαμπέλ Τόμας αντικατέστησε την κυρία Τροτμάν ως τακτικό μέλος της Επιτροπής. Την καλωσορίζουμε. Επίσης ο κύριος Ζανλουί Κοτινή αντικατεστά την κυρία Γκρελιέ ως αναπληρωματικό μέλος. Σας καλωσορίζουμε και εσάς στην Επιτροπή μας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Ανταλλαγή απόψε με τον κύριο Πασκάλ Σαμπουρέ, Διευθυντή της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλίας στο Βίγκο. Να καλωσορίσουμε τον Διευθυντή, ο οποίος θα μας ε, παρουσιάσει την έκθεση για τα πέντε χρόνια εργασίας ε, του οργανισμού και θα μας παρουσιάσει και τις, ε, το μελλοντικό έργο. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ και ξέρετε ότι θα σας την ε, επιστρέψουμε κατά κάποιο τρόπο την επίσκεψη αυτή ερχόμενη εμείς στο Βίγκο. Σας δίνω το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που δίνετε τη δυνατότητα στον ε, Οργανισμό Ελέγχου της Αλληλείας να δώσει κάποιες πληροφορίες όσον αφορά τις δραστηριότητες των εργασιών μας και του προγράμματος μέχρι το Μάρτιο. Τον Οκτώβριο θα γίνει μια νέα παρουσίαση που θα σας παρουσιάσει τις υπόλοιπε δραστηριότητες και αυτές που είναι ακόμα ανεξέλιξη. Αν μου επιτρέπετε θα αλλάξω θέση για να πάω κοντά σε έναν υπολογιστή. Euh, Καταρχήν θα ήθελα να σας παρουσιάσω τρία συγκεκριμένα κεφάλαια. Το θέμα της διακυβέρνησης, πενταετής αξιολόγηση, συστάσεις οι οποίες έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκαν από αυτό το Συμβούλιο στο τέλος της αξιολόγησης και του σεμιναρίου που έλαβε χώρα στις 14 Μαρτίου του 2012, καθώς και το σχέδιο εργασιών, πρόγραμμα εργασιών για το 2013 και το πολιετές 2013-2017. Κατόπιν αν μας μείνει χρόνος, θα κάνω μία παρουσίαση των ενεξελίξη δραστηριοτήτων και βεβαίως το τι θα μπορούσαμε να αναλάβουμε στο μέλλον. Η αξιολόγηση έγινε βάσει του άρθρου 39 του κανονισμού, του ιδρυτικού κανονισμού της ε, υπηρεσίας του οργανισμού και τα πέντε πρώτα χρόνια ύπαρξης ε, αυτού του φορέα έγινε η πρώτη αξιολόγηση όσον αφορά την λειτουργία του οργανισμού μας. Αυτό έγινε από διάφορες ε, εταιρείες. Όπως καταλαβαίνετε δεν πρόκειται να, τους, ε, να αναφέρω τα ονόματά τους για κατανοητούς λόγους. 85.000 ευρώ είναι το κόστος. Η αξιολόγηση αυτή είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ αποτελεσματική και χρήσιμη για μας. Το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης είναι ότι εργαστήκαμε με αποτελεσματικό τρόπο, η διακυβέρνηση ήταν ε, σωστή, τα αποτελέσματα αξιόλογα. Βεβαίως, μπορούμε ακόμα να βελτιωθούμε και η αρχή αξιολόγησης θεωρεί ότι όσον αφορά τα αποτελέσματά μας και βάσει πολύ συγκεκριμένων κριτηρίων, αποτελεσματικότητας, βιωσιμότητας, ε, η εργασία του οργανισμού θεωρείται αποτελεσματική και ε, ελπιδοφόρα. Πρόκειται βεβαίως για μια λειτουργία σε ένα πάρα πολύ τεταμένο δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Εδώ βλέπετε τι ε, μπορεί κανείς να διαβάσει στο άρθρο 116 της ε, έκθεσης. Από την 1η ε, Ιανουαρίου του 2012 αλλάξαμε όνομα Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αλίας. Η δραστηριότητά μας στηρίζεται σε τρεις κατευθυντήριες γραμμές, σε τρεις άξονες. Καταρχήν η εργασία των αξιολογητών, του Διοικητικού Συμβουλίου, των κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ελεγκτικού Συνεδρίου, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλοι φορείς με τους οποίους έχει ο οργανισμός μας επαφές, όπως η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκός Οργανισμός ε, Ασφάλειας ε, τη Θάλασσα, καθώς και η Frontex. Και άλλοι μη κυβερνητικοί οργανισμοί και περιφερειακοί οργανισμοί. Όλη αυτή η ανάλυση έχει σαν αποτέλεσμα ότι το 76% προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τα κράτη-μέλη και κατόπιν 20% από τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Η έκθεση αξιολόγησης αυτή καθεαυτή βασίζεται, όπως σας είπα, σε τρεις άξονες. Είναι ένα τρίπτυχο. Μιλήσαμε για τη διακυβέρνηση, την αποτελεσματικότητα και για να είμαι σύντομος θα σας κάνω μια παρουσίαση πολύ συγκεκριμένη την πτυχή της ε, ε, αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και όσον αφορά τα συμπεράσματα της αξιολόγησης για τη διακυβέρνηση θα τα αναφέρω μόνο στα συμπεράσματα και στις συστάσεις που γίνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, θα μιλήσουμε για την απόδοση, για την αποτελεσματικότητα, για την αηφορία. Όταν σας μιλάω για αηφορία ή βιωσιμότητα, δεν αναφέρομαι στους πόρους βεβαίως, αλλά στην εργασία του οργανισμού, στις δυνατότητες που διαθέτει, έτσι ώστε να έχει θετική επίπτωση την ε, ενιαία μέθοδο που χρησιμοποιείται όσον αφορά τους ευρωπαϊκούς ελέγχους. Τώρα, όσον αφορά το ακριβές ε, της εργασίας αυτής, ο αξιολογητής θεωρεί εδώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο επιχειρησιακός συντονισμός και την ίδια ώρα θεωρεί ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς, δηλαδή τα κράτη-μέλη, είναι διατεθειμένα να ξεπεράσουν τη σημερινή τους δράση και να δεσμευθούν σε μια περιφερειακή δράση ασχολούμενη πολύ περισσότερο και εμπλεκόμενη σε περιφερειακά σχέδια και σε μια συνεχή δράση. Δεύτερη διαπίστωση όσον αφορά την ανάπτυξη των ε, δυνατοτήτων όσον αφορά παραδείγματο χάρη την κατάρτιση, τα συστήματα πληροφορικής. Η αξιολογήση θεωρεί εδώ ότι είναι πολύ σωστή η δράση Είναι όμως λιγότερο πεπισμένη η αξιολογική, η αξιολογική αρχή όσον αφορά τα αποτελέσματα αυτής της ε, πτυχής. Δηλαδή, δεν υπάρχει εδώ αρκετό συντονισμός στις διάφορες αλευτικές ε, περιφέρειες, περιοχές. Και μπορείτε να δείτε σε αυτή τη γραφική παράσταση τα διάφορα σχέδια κοινή δραστηριότητας και την καταπολέμηση της παράνομης αλίας σε γενικές γραμμές βλέπετε ότι είναι ικανοποιητικά τα αποτελέσματα πάνω από 80% δηλαδή των αποτελεσμάτων. Βλέπετε εδώ για τη Μεσόγειο, για τον τόνο, Βόρειος Ατλαντικός επίσης 80%. Για τη Βόρεια Θάλασσα και τις δυτικές περιοχές και τη Βαλτική. Για το IUU, επίσης βλέπετε, αποτελέσματα είναι εξαιρετικά ικανοποιητικά πάνω από 90%, δηλαδή κατά πολέμηση της παράνομης αλίας. Όταν εξετάσουμε τις δυνατότητες, η δραστηριότητα εδώ είναι βεβαίως και πιο καινούρια αλλά και τα αποτελέσματα λιγότερο, απο, λιγότερο θετικά. Εδώ θα έλεγα ότι υπάρχει πρώτον θέμα χρηματοδότησης. Ε, έχει ενσωματωθεί αυτή η δραστηριότητα πολύ πρόσφατα στις ε, ευρωπαϊκές ε, δραστηριότητες. Ο έλεγχος ξεκίνησε με τον κανονισμό 404 που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2011. Όσον αφορά το Core την κατάρτιση, βλέπετε εδώ ότι δημιουργήθηκε ένα επιχειρησιακό κέντρο στον οργανισμό. Επίσης, εξαγορά ενός σκάφους ναυλωμένου και το fishnet, το δίκτυο. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του οργανισμού της δράσης μας, η έκθεση θεωρεί ότι όσον αφορά την διοικητική και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα είχαμε πολύ θετικά αποτελέσματα. Πολύ σύντομα δηλαδή ο οργανισμός δημιούργησε πολύ ισχυρούς δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράφηκαν συμβάσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η συνεργασία με άλλους φορείς και οργανισμούς ήταν εξαιρετική, όπως παραδείγματο χάρη με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θαλάσσιας Ασφάλειας. Το Βασίλειο της Ισπανίας επίσης, με το οποίο έχουμε εξαιρετικές σχέσεις. Παρ' όλα αυτά, η αξιολόγηση αναφέρει ότι επηρεάζεται η, επιχειρησιακή συγγνώμη, αποτελεσματικότητα από το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια περιφερειακή και απομακρυσμένη περιοχή, κόστος δηλαδή, εξαιτίας ε, της ε, εγκατάστασής μας και βεβαίως και κάποιες άλλε ανησυχίε όσον αφορά τη βιομάζα για τον κόκκινο τόνο και όσον αφορά την μεταφορά του από τον τόπο αλίας ε, στην μεταφορά. Και βεβαίως οι δυνατότητες αυτές, όπως σας είπα, έχουν αναπτυχθεί με βραδύτερους ρυθμούς, κάτι το οποίο αναφέρεται στην έκθεση. Όσον αφορά το θέμα των δυνατοτήτων, εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολο να χρησιμοποιήσει κανείς συγκεκριμένους δείκτες. Γιατί βεβαίως εδώ παίζει ρόλο ο συντονισμός, η αποτελεσματικότητα του συντονισμού που εδώ εμπίπτει στο προηγούμενο κεφάλαιο και βεβαίως υπάρχουν παράμετροι όπως η αμοιβαία εμπιστοσύνη, η οικονομική απόδοση και βεβαίως η συμβατότητα. Σήμερα μπορεί να πει κανείς ότι είναι πολύ δύσκολο να αποδώσει κανείς στον επιχειρησιακό συντονισμό τη βελτίωση της συμβατότητας αυτές τις αλλιευτικές ε, περιφέρειες. Υπάρχει το θέμα των κυρώσεων και υπάρχει το θέμα της μείωσης της απόδοσης. Παρ' όλα αυτά, τα κράτη-μέλη καλούνται εδώ, όπως και ο οργανισμός, να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Ο οργανισμός παίζει ένα ρόλο συντονισμού για τη βελτίωση της συμμόρφωσης. Όσον αφορά λοιπόν την αποτελεσματικότητα, θα πρέπει να κοιτάξουμε προσεκτικές παρατηρήσεις το σχέδιο του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δραστηριότητα του οργανισμού μας. Βελτιώσαμε την εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών, την πολυμερή συνεργασία, τη διμερή συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών ε, μεταξύ των κρατών μετών μελών και βεβαίως αποφύγαμε επικαλύψεις και βελτιώσαμε την συνέργεια, ε, τη συνεργασία όσον αφορά τους ελέγχους. Δημιουργήσαμε διμερείς σχέσεις για ελέγχους και όσον αφορά τη μείωση του κόστους Βεβαίω, εδώ υπάρχουν πολλέ διαφορετικέ ε, απόψεις μεταξύ των κρατών μελών, γι' αυτό και βασιζόμαστε σε διμερείς ε, επαφές και συμφωνίες. Για τον περιορισμό του κόστους βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ θετική η προσέγγιση του Διοικητικού Συμβουλίου και εδώ βλέπετε ότι ε, συμφωνούμε με την έκθεση αξιολόγησης και αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ θετικό. Όσον αφορά τις ε, επιπτώσεις, πάρα πολύ σημαντική είναι εδώ η βελτίωση των ε, επιπέδων των αποθεμάτων. Είναι ένα θέμα για το οποίο θεωρούμε ότι ο οργανισμός έχει συμβάλει θετικά. Η αξιολόγηση εδώ δεν ε, αντιμετωπίστηκε από τα κράτη-μέλη με πολύ αποφασιστικό τρόπο. Υπήρξε δηλαδή λίγο θέμα πρόσβαση στα δεδομένα σε κάποιες περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, βελτιώθηκε η κατάσταση των αποθεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παραδείγματο χάρη στη Βαλτική. Και εδώ ο ρόλος του οργανισμού είναι καθοριστικός. Όσον αφορά την αηφορία των μεθόδων που χρησιμοποιεί ο οργανισμός, πρέπει να σας πω ότι η θέση της αρχής αξιολόγησης είναι πάρα πολύ θετική. Υπογραμμίζει βεβαίως ότι πρέπει να υπάρξουν επίσημες συμφωνίες, συνεργασίας, κάτι που δεν υπάρχει πάντα και ίσως έτσι θεωρεί η αξιολόγηση, είναι πολύ νωρίς για να γίνει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση της ε, βιωσιμότητας. Και βεβαίως αυτά απευθύνονται και στο Διοικητικό Συμβούλιο. 14 Μαρτίου οργανώθηκε ένα σεμινάριο στο Βίγκο. Εκεί υπογραμμίστηκαν τα αδύναμα σημεία, τα θετικά σημεία της στρατηγικής του οργανισμού και προετοιμάστηκε η στρατηγική του μέλλοντος. Όλα αυτά πρέπει να σας πω ότι εγκρίθηκαν την επομένη από το Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε με λεπτομέρεια όλες αυτές τις συστάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρόκειται για την στρατηγική του οργανισμού, για, τα, για το μέλλον και βεβαίως θα ενσωματωθούν στο πρόγραμμα εργασιών του οργανισμού. Πρώτη σύσταση, πρώτη διαπίστωση. Το Level Planning Field και η συμμόρφωση πρόκειται για τους δύο στόχους, μακροπρόθεσμους αλλά και άμεσους στόχους για τον οργανισμό. Περιφερειακή προσέγγιση, καθώς και κοινά σχέδια μακροπρόθεσμα και συνεχή, και αυτό είναι κάτι το οποίο το είδε με πάρα πολύ θετικό τρόπο το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο όμως βεβαίως υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρξει νομική βάση και να θεσπιστούν και προτεραιότητες όσον αφορά τα είδη. Εδώ η θέσπιση και ο καθορισμός προτεραιοτήτων, καθώς και η αξιολόγηση του ρόλου του οργανισμού βάσει της αρχής της βέλτιστης μεθόδου για την προστιθέμενη αξία καθώς και την επιλογή στρατηγικών εναλλακτικών από τη στιγμή που αλλάζουν οι προτεραιότητες σε μια συγκεκριμένη περιοχή και δεν υπάρχει ε, προτεραιότητα για ένα συγκεκριμένο είδος στην περιοχή αυτή. Ο δικός ε, χάρτης για κάποιες συγκεκριμένες περιοχές ε, όσον αφορά το core curricula, την κατάρτιση και αυτό είναι κάτι το οποίο το υπογραμμίζει και η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημιουργία προγράμματος εργασίας όσον αφορά το περιφερειακό επίπεδο για παρατηρητές και για επιθεωρητές από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας και ανάπτυξη δικτών για το capacity building και την μέτρησή του. Πρόκειται για ένα σύστημα ελέγχου, πρέπει να γίνει η μέτρηση της οικονομικής αποτελεσματικότητας αυτής της μεθόδου και βεβαίως να ληφθούν υπόψη και στοιχεία δημοσιονομικά από μέρους όλων των κρατών μελών. Προτείνεται επίσης ο οργανισμός να ενημερώσει για τις βέλτιστες πρακτικές σε επίπεδο διοικητικής συνεργασίας, αποτελεσματικότητας, να ενσωματώσει στα προγράμματά της ανάλυση κινδύνου και βεβαίως εδώ υπάρχει και η επιστημονική συμβουλή όσον αφορά τα αποθέματα των διαφόρων περιοχών. Επίσης, ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του οργανισμού και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διευκρινίζοντας την αξιοπιστία των δεδομένων. Αυτό είναι κάτι που συνδέεται άμεσα με τον κανονισμό για τον έλεγχο και βάση βεβαίως της συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς όπως προβλέπει και ο κανονισμός. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης υιοθετεί την σύσταση να ε, επιστήσει στην προσοχή σε στρατηγικά θέματα. Και αυτό βάσει της γραπτής διαδικασίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί επίσης ότι θα πρέπει να σκεφτεί και το άνοιγμα σε άλλους ε, φορείς. Να υπάρχει δηλαδή μία εκπροσώπηση και άλλων φορέων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι είναι πολύ νωρίς έτσι ώστε να τροποποιηθεί ο κανονισμός και παρόλα αυτά θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα οδηγός, ένα εγχειρίδιο όσον αφορά τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών. Αυτά όσον αφορά την πενταετή αξιολόγηση, την αξιολόγηση του πενταετούς προγράμματος, της πενταετούς λειτουργίας του οργανισμού, με σκοπό βεβαίως να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά μας, την απόδοσή μας και την δημοσιονομική λειτουργία του οργανισμού. Από εδώ και πέρα θα σας ε, παρουσιάσω το πρόγραμμα εργασιών του οργανισμού, τις ε, προτεραιότητες και βεβαίως το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει επίσης να πάρει και κάποια μέτρα περιοριστικά. Δεν μπορώ να προβλέψω ποιες θα είναι αυτές οι προτεραιότητες. Και όσον αφορά τη δραστηριότητα του οργανισμού, όπως σας είπα, θα βασιστούμε σε τρεις κατευθυντήριες γραμμές Σιακικός συντονισμός και συνεργασία, συνεργασία με τα κράτη-μέλη, με τις τρίτες χώρες και βεβαίως η ανάπτυξη των δυνατοτήτων. Όσον αφορά Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο θα υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο στις 9 και 10 Οκτωβρίου, προτείνουμε να υπάρξει μια περιφερειακή προσέγγιση. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να προτρέξουμε της κοινή αλλιευτικής πολιτικής. Και όσον αφορά το σύνολο των ε, περιοχών στηριοποιούμαστε, υπάρχει και η Μαύρη Θάλασσα, καθότι ο οργανισμός έχει συνάψει μια συμφωνία ελέγχου με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία με σκοπό να υπάρξει συντονισμός ε, για τη Βόρεια Θάλασσα, για την Μαύρη Θάλασσα, συγγνώμη. Αξιολόγηση λοιπόν των επιπτώσεων όσον αφορά τους ελέγχους που διενεργούνται και η ανάλυση κινδύνου. σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των δυνατοτήτων και έχοντα υπόψη μα και τον προπολογισμό σήμερα, είναι ζωτική σημασία για τον οργανισμό αλλά και για όλα τα κράτη-μέλη, θα έλεγα. Η ανάπτυξη συστημάτων πληροφοριών, βέβαια, πάντοτε ε, με πλήρη σεβασμό στου κανόνε και τη ε, ιδιωτική ζωή, όπω προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Αυτό είναι και ο ρόλο του επόπτη των ε, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Χρειάζονται όμως τα συστήματα πληροφοριών για την ε, καθημερινή εργασία. Το ΕΡΕΣ λοιπόν, ε, το, book, το ηλεκτρονικό βιβλίο, το σύστημα επίσης ανταλλαγής ε, πληροφοριών για να μπορεί ένα επιχειρησιακό κέντρο εικονικά να μπορεί να μεταφερθεί όπου και αν βρίσκεται το συντονιστικό κέντρο. Υπάρχει επίσης το JATE, που είναι ένα πρόγραμμα για τον σχεδιασμό των μέσων ελέγχου, αν υπάρχει ένα σχέδιο κοινή ανάπτυξης. Υπάρχει επίσης εκπαιδευτική πλατφόρμα, καθώς και ένα σχέδιο το οποίο λέγεται η IR στα αγγλικά, ε, που είναι ένα σχέδιο για τις ε, εκθέσεις ελέγχου, δηλαδή προβλέπει την ανταλλαγή ε, στοιχείων όταν υπάρχει επιθεώρηση πλοίων. Ο οργανισμός θα μπορούσε λοιπόν να αναπτύξει το εν λόγω πρόγραμμα για όλα τα κράτη-μέλη, τέλος πάντων για όσοι ενδιαφέρονται, ώστε να μειωθεί το κόστος ανάπτυξης του προγράμματος. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών ε, και των επιθεωρητών. Είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο αυτό. Αρχικά έχουμε τον έλεγχο στη θάλασσα, το πρώτο σκέλος. Περιμένουμε να είναι έτοιμο το Φεβρουάριο του 2013. Επίσης, ε, η παροχή βοήθεια στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα ακόμη σημαντικό σκέλο για την υλοποίηση της ε, αναφερμένη πολιτικής αλίας. Παραδείγματο χάρη, συμβάλλουμε στον προβληματισμό που γίνεται για διάφορα θέματα τα οποία προκύπτουν. Νέες τεχνολογίες επίσης για τη μείωση του κόστους του ελέγχου χρησιμοποιώντας τα δορυφορικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι ένα σχέδιο αυτό το οποίο ήδη αποτέλεσε αντικείμενο πιλωτικού προγράμματος που ολοκληρώνεται ως ονούπο και νομίζουμε ότι θα μπορούσε να είναι επιχειρησιακό, να βρει εφαρμογές δηλαδή πρακτικές τους επόμενους μήνες ή χρόνια αν το ΔΣ θεωρήσει ότι αυτό θα ήταν θετικό για τον έλεγχο. Η συνεργασία επίσης με τρίτες χώρες κατόπιν αιτήματος της Κομισιόν ε, δεν είναι ένας τομέας ε, που από μόνη της αναλαμβάνει πρωτοβουλία υπηρεσία μας. Οι δυνατότητες ε, συνεργασίας μέχρι στιγμής αναπτύσσονται με τον Καναδά και τις χώρες της νότιας όχθης της Μεσογείου σε ό,τι αφορά τον ερυθρό τόνο συγκεκριμένα. Είχαμε και ένα σεμινάριο που οργανώσαμε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν από 10 ημέρες στο Βίγκο έλαβαν σε αυτό το σεμινάριο σχεδόν μέλος, μέρος σχεδόν όλες οι χώρες της Μεσογείου. και με την Νορβηγία επίση θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε και τι νήσου Φερόση γιατί όχι και την Ισλανδία στο πλαίσιο τη εργασία μα με τον Βόρειο Ατλαντικό. Ο Καναδά είναι πολύ σημαντική χώρα εταίρο στο πλαίσιο του ΝΑΦΟ. Όπω και η ΙΠΑ ε, στον ε, τομέα τη καταπολέμηση ε, τη παράνομη αλία. Προπολογισμό του 2013 τον γνωρίζετε ουσιαστικά πρόκειται για τον προπολογισμό που ενέκρινε το ΔΣ όταν συνεδρίασε στις 15 Μαρτίου του 2012 είναι ένας προϋπολογισμός ε, που μετά την πρόταση του Συμβουλίου επηρεάστηκε κατά 73 ε, εκατομμύρια προτείνει στον τίτλο 1 και στον ε, τίτλο 2 μείωση το Συμβούλιο. Στο, κατά το έτος 2012 ήταν αρκετά υψηλή, πολύ υψηλή εκτέλεση του προϋπολογισμού. Κατά το 99% εκτελέστηκε ο προϋπολογισμός, όπως βλέπετε και στο γράφημα αυτό. Τώρα, πολύ γρήγορα θα ήθελα να σας αναφέρω τα επιχειρησιακά. Τι έγινε δηλαδή κατά τη διάρκεια του 2012 στο πρώτο εξάμεινο ε, του, του 12 και επίσης και τι έγινε στο 2011. Ο οργανισμός μας συντόνισε μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2012 5.295 επιθεωρήσεις Είχαμε 332 σοβαρές υποθέσεις επιθεώρησης μεταξύ αυτών. Βλέπετε στον πίνακα τα σχετικά στοιχεία. Οι περισσότερες παραβάσεις αφορούν ε, την δήλωση των αλευμάτων ουσιαστικά. Σε κάποιες περιπτώσεις βέβαια είναι πολύπλοκη η δήλωση των ε, αλευμάτων, όπως για τον τόνο για παράδειγμα, αλλά είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό, πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ε, δημιουργεί προβλήματα στον ε, ληφτικό στόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολή στοιχείων. Πιστεύουμε ότι με το ηλεκτρονικό σύστημα αυτού του είδους οι συστημικές παραβάσεις θα μειωθούν. Σε αυτό το γράφημα, σε αυτή τη γραφική παράσταση βλέπετε το ποσοστό των παραβάσεων σε σχέση με το σύνολο των επιθεωρήσεων που έγιναν. Δεν είναι γραμμικά ε, τα στοιχεία αυτά, έξω και πρέπει με προσοχή να, να δούμε ε, τα στοιχεία για την εξέλιξη που είχαμε το 2012 γιατί αφορούν μόνο το πρώτο εξάμεινο το 2012. Βέβαια, σε ό,τι αφορά τις περισσότερες περιπτώσεις πλήν της Βαλτικής, βλέπουμε μείωση του ποσοστού αυτού παραβάσεων. Αυτό είναι ενθαρρυντικό βέβαια. Καλό θα είναι βέβαια να δούμε πρώτα πώς θα εξελιχθεί συνολικά το έτος 2012. Εδώ βλέπετε μια άλλη γραφική παράσταση. Το 2011 ο οργανισμός μας ειτώνησε σχεδόν 10.000 επιθεωρήσεις. Στη θάλασσα ήταν σχεδόν οι 2.200 από αυτές. Και πάλι δεν έχουμε τα οριστικά στοιχεία, επαναλαμβάνω, για το 2012, γιατί είμαστε ακόμη στο πρώτο εξάμεινο. Βλέπετε όμως ότι στο 2012 ο αριθμός των επιθεωρήσεων στη θάλασσα έχει ήδη φτάσει ε, σχεδόν το συνολικό αριθμό των επιθεωρήσεων στη θάλασσα του 11, άρα έχουμε αύξηση των επιθεωρήσεων. Ιδίως στα δυτικά ύδατα στα μικρά πελάγια και στην Βαλτική για το Σολομό θα γίνει μια ειδική δραστηριότητα και έτσι θα έχουμε και τα στοιχεία σύντομα να τα συμπεριλάβουμε σε αυτή τη γραφική παράσταση και για τη Βαλτική. Για τον τόνο, τον ερθινό τόνο το 2012 βλέπετε εδώ κάποια στοιχεία. Σημαντικά τα μέσα τα οποία αναπτύχθηκαν αλλά το σκάφος το οποίο είχαμε αναβλώσει από την 1η Απριλίου του 12 και μετά δεν είναι αναβλωμένο, άρα δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει. Βλέπετε πάντως τα στοιχεία αυτά και σε σχέση με τις ε, περιπολίες. Πόσα σκάφη λοιπόν επιθεωρήθηκαν. Δεν έχει λήξει βέβαια η εποχή αλλία του Ριθρουτών ακόμη. Μέχρι 15 Οκτωβρίου μπορεί να διατηρηθεί, ίσως και μέχρι το τέλος του χρόνου σε κάποιες περιπτώσεις. Έχουμε επιθεωρήσει μέχρι τώρα 372 σκάφη. 33 παραβάσεις διαπιστώθηκαν. Και αφορούσαν κυρίως τις δηλώσεις αλλιευμάτων. Ή τα έγγραφα, τα σχετικά με τα αλλιεύματα, το ε, ημερολόγιο και έχουμε δει και κάποιες διαφορές σε σχέση με, την, ε, με τα βίντεο, γιατί ξέρετε ότι βιντεοσκοπείται η δραστηριότητα. Ε, πώς τώρα μπορούμε να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας με τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Για τον ερθροτόνο κάναμε μία προσπάθεια να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τα δεδομένα τα οποία έχουμε, VMS, ε, AIS ή τα δορυφορικά, τι πληροφορίες μπορούμε να συλλέξουμε για την γενικότερη δραστηριότητα των σκαφών. Έχουμε και το IES που είναι αυτόματη συλλογή δεδομένων, τα οποία στοιχεία δίνουν τα, και τα εμπορικά πλοία, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό. Έχουμε και IS τα ε, στοιχεία του οποίου λέγονται μέσω δορυφόρου, Έχουμε και τα sightings, δηλαδή την αναγνώριση ε, πλοίων. Βλέπετε ένα χάρτη εδώ που βλέπετε το σύνολο των διαθέσιμων πληροφοριών. Και με τη διασταύρωση των στοιχείων μπορούμε να ε, συλλέξουμε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τις συμπεριφορές. Εδώ βλέπετε μια κανονική δραστηριότητα τον Ιούνιο στα νότια της Σικελίας. Γύρω στη Μάλτα βλέπετε ότι επικεντρώνεται κυρίως η δραστηριότητα. Βλέπουμε βέβαια και κάποια λεφτικά σκάφη που δεν τα είχαμε ε, αλλιές και κάποια άλλα εμπορικά πλοία, των οποίων είναι και κάποια ε, πλοία ψυγεία που δεν έχουν θέση σε λειτουργία το σύστημα VMS. Τι βλέπουμε εδώ. Εδώ εντοπίσαμε ένα πλοίο, ένα σκάφος, που φαινόταν να μην έχει άδεια ICAT. Κάναμε λοιπόν διασταύρωση των στοιχείων μας από βάση δεδομένων με τα δεδομένα VMS. Μόνο ο διαχειρός μπορούσε να αποκτηθεί σχετική πληροφορία μέχρι τώρα, αλλά τώρα με την αυτοματοποίηση που έχουμε μπορούμε να εντοπίσουμε την παρουσία όλων των πλοίων, όλων των σκαφών και να διαπιστώσουμε κατά πόσο έχουν όχι όλες τις σχετικές απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες και μπορούν, αν έχουν βέβαια την άδεια VMS, τα σκάφη να λιεύουν ομίμω. Εδώ μια άλλη περίπτωση. Έχουμε ένα λευτικό πλοίο που διαθέτει VMS και ένα άλλο που δεν έχει VMS, αλλά έχει το AIS. Άρα με βάση τα δεδομένα του AIS μπορούμε να δούμε τις δραστηριότητες αυτού του σκάφους, τέλος πάντων να ε, συγκεντρώσουμε πληροφορίες για την παρουσία, το λόγο της παρουσίας του στην περιοχή αυτή. Μια άλλη δραστηριότητα, πάλι παράδειγμα, ένα λευτικό σκάφος από τη Ρωσία το οποίο ε, μέσα στη Μεσόγειο το παρακολουθήσαμε, βλέπετε την πορεία του. Ε, υπήρξε κάποια ανησυχία την παρουσία αυτού του σκάφους. Ε, χάρη λοιπόν σε αυτό το σύστημα καταφέραμε κάνοντας πάλι διασταύρωση στοιχείων να διαπιστώσουμε ότι δεν υπήρξε καμία ούτε αλληλευτική ούτε εκφορτική δραστηριότητα από αυτό το σκάφος. Δεν σταμάτησε καθόλου. Και διαπιστώσαμε και όλη του την διαδρομή με τα διάφορα δεδομένα που έχουμε. Κάναμε λοιπόν τη σχετική διασταύρωση των στοιχείων και είδαμε και τη μέση του ταχύτητα που μας έδειχνε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να άσκησε κάποια άλλη ε, δραστηριότητα λόγω της ταχύτητας που είχε. Θα έχουμε λοιπόν και το πρόγραμμα εργασίας τώρα. Για τι επιχειρησιακές μα δραστηριότητε, να πω και κάτι. Τι μπορεί να γίνει στο μέλλον τον οργανισμό. Θα σας δώσω κάποιες, ε, κάποια στοιχεία. Έχουμε τη μεταρρύθμιση ε, του ελέγχου και της κοινή αλληλευτική πολιτική. Σήμερα είναι σημαντικό ότι τα κράτη-μέλη ζητούν από τον οργανισμό να στηρίξει πολύ περισσότερο ε, τον έλεγχο και όχι μόνο το συντονισμό, τον επιχειρησιακό συντονισμό. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι μια άποψη που την ε, ακούμε συχνά και σε επίπεδο ΔΣ. Μια άλλη σημαντική πτυχή είναι η συμβολή που θα μπορούσε να έχει ο οργανισμός μας στο πλαίσιο των νέων διατάξεων της κοινή αλληλευτικής πολιτικής όταν θα έχει ε, τροποποιηθεί και δει συμμετοχή του οργανισμού σε κάποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες και στην εκπόνηση των μεθόδων ελέγχου. Ιδίως σε ό,τι αφορά την απαγόρευση των απορρίψεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα θα πρέπει να ορίσει έναν οργανισμό για την ε, συλλογή των δεδομένων και νομίζω ότι θα μπορούσε ο δικό μα οργανισμό να είναι αυτό ο οργανισμό ιδίω για ένα μέρο των στοιχείων. Επίση θα πρέπει τα κράτη-μέλη να βοηθηθούν για να δημιουργήσουν, ε, είπαμε, συστήματα πληροφοριών. Και αυτό θα είναι μια νέα μορφή συντονισμού. Γιατί το κόστο ανάπτυξη ενό συστήματο πληροφοριών, να σα επισημαίνω ότι είναι υψηλό. Αν τα κράτη-μέλη, τα 20 κράτη-μέλη ή με την Κροατία τα 21 αναπτύσσουν το καθένα ξεχωριστά ένα σύστημα πληροφόρων που δεν θα είναι και κατά ανάγκη ταυτόσουμε με τα άλλα, εδώ καταλαβαίνετε ότι υπάρχει κίνδυνο να δημιουργηθεί πολύ σημαντικό κόστο. Και δεν είναι και η καλύτερη συνέργεια σε επιχειρησιακό επίπεδο. Εξού και ο οργανισμό θα μπορούσε να εκπονήσει, να καταρτήσει συστήματα για όλα τα κράτη-μέλη. Και τέλος, ο οργανισμός θα μπορούσε να συνεισφέρει περισσότερο στη νέα προσέγγιση μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ειδικά προγράμματα ελέγχου και επιθεώρησης. Σήμερα η κοινή πολιτική ε, αλληλίας θα μπορούσε να έχει μια προσέγγιση όλο και περισσότερο προσανατολισμένη στα αποτελέσματα με τη δημιουργία ενός συστήματος αξιολόγησης με ένα επίπεδο στρατηγικής και ένα επίπεδο τακτικής. Στο επίπεδο της συνεργασίας υπάρχουν αυτά τα δύο επίπεδα στο επίπεδο του οργανισμού μας. Για την ανάπτυξη ενός κοινού προγράμματος έχουμε το στρατηγικό επίπεδο που είναι η λεγόμενη Διευθύνουσα Επιτροπή και έχουμε και την κοινή ομάδα τακτικής που είναι το δεύτερο επίπεδο. Αυτή η προσέγγιση θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε μια καλύτερη ανάλυση τόσο του κόστους όσο και των αποτελεσμάτων. Και αυτά θα μπορούν να ελεγχθούν και να μετρηθούν. Θα μπορούμε επίσης να ορίζουμε στόχους, ποσοστά παραβάσεων, πόσο θέλουμε να μειωθούν δηλαδή οι παραβάσεις και έπειτα να μετρούμε. Έχουμε τα μέσα για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς και να αξιολογούμε βέβαια το κόστος και το αποτέλεσμα. Εδώ είναι ένα παράδειγμα του input. Αριθμός επιθεωρήσεων, μέρο στη θάλασσα, επαλήθευση αξιολόγησης ε, και ε, εκτίμηση του κόστους και του αριθμού των παραβάσεων. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ. Μακρηγόρησα λιγάκι. Ε, ζητώ συγγνώμη, αλλά με παθιάζει αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Δύο μόνο συνάδελφοι ζουν το λόγο. Τρεις. Λοιπόν, καλώς. Θα πάρω το λόγο τέσσερις, τέσσερις συνολικά. Η κυρία Γκαρθία Γέρο. Καλημέρα σας, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ που είναι το λόγο, κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής. Πρώτα απ' όλα, να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον Διευθυντή του οργανισμού για τις λεπτομερείς αυτές τις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης και, και την έκθεση αξιολόγησης των πέντε ετών ζωής του οργανισμού. Ο απολογισμός είναι θετικός, σύμφωνα με τα λεγόμενά σας, και εγώ δεν τον πισβητώ καθόλου. Υπάρχουν όμως κάποια θέματα στα οποία αναφερθήκατε, και επιθυμώ να θέσω κάποιες ερωτήσεις για να μας εξηγήσετε καλύτερα ακριβώς ότι σε τι συνίσταται οι εργασίες του οργανισμού και σε ποιο βαθμό υπάρχει συνέχεια σε αυτές τις εργασίες. Κάτι άλλο τώρα. Πώς γίνεται η συνεργασία όλων των κρατών μελών του οργανισμού ως η συνεργασία είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση και τον συντονισμό των δεδομένων, ώστε να έχουμε επιθεωρήσει πρακτικά να αντιμετωπίσουμε την αλία IUU, την παράνομη λαθρέα και άναρχη αλία. Υπάρχει συνεργασία πρακτικά, ναι ή όχι. Θα πρέπει εμείς εδώ να γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί που δεν συνεργάζονται. Γιατί αλλιώς πώς θα επιτύχουμε αυτό τον τόσο ε, θεμελιώδη στόχο για την αντιμετώπιση της αλληλείας IUU. Επίσης, αν έχω καταλάβει καλά, ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη συλλογή και χρησιμοποίηση αυτών των δεδομένων και ώστε να κάνει και επιθεωρήσεις στην ανοιχτή θάλασσα, χρειάζεστε ένα σκάφος και υπάρχει το πρόβλημα βεβαίω τη περικοπή του προπολογισμού λόγω τη κρίση και τελικά δεν θα έχετε την να χρησιμοποιείτε αυτό το, το σκάφο. Κατάλαβα καλά ή ε, τα έχω μπερδέψει. Ε, αν είναι αλήθεια αυτό που λέω, είναι πολύ δύσκολη παρακολούθηση στην ανοιχτή θάλασσα για τον εντοπισμό σκαφών όπως εκείνου του ρωσικού σκάφους ε, που γνωρίζουμε. Εγώ εξ όσων γνωρίζω δεν έχει γίνει κάτι συγκεκριμένα. Σε σχέση με τον προπολογισμό, είναι τελευταίο σχόλιο για αυτά τα δύο project που αναφέρατε. Κατ' εμέ, αυτό που βλέπω, η δική μου άποψη είναι μία οπισθοχώρηση. Βήματα πίσω σε σχέση με δραστηριότητες που θα πρέπει να φέρει πέρα ο οργανισμός. Αυτή είναι η δική μου ταπεινή γνώμη τουλάχιστον. Δηλαδή τα κράτη-μέλη δεν αρκούν από μόνα τους να φέρουν εις πέρας αυτούς τους ελέγχους. Χρειάζεται και ένας έλεγχος επιθεώρησης σε ανανότερο επίπεδο ή τουλάχιστον ε, ο οργανισμός, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνουν αυτόν τον υπερεθνικό έλεγχο. Με βάση τους οικονομικούς πόρους που διαθέτεται, η αλήθεια είναι ότι εγώ γνωρίζω ότι κάνετε εξαιρετική δουλειά. Και στο μέτρο των δυνατών που έχουμε και εμείς ως Ευρωβουλευτές πρέπει να σας υποστηρίξουμε ώστε να συνεχίζετε να έχετε τους κατάλληλους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, ώστε να συνεχίζετε να εμβαθύνετε σε αυτές τις τόσο σημαντικές δραστηριότητε. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ οι υπόλοιποι ε, αγορητές να είναι πιο συνοπτικοί στις ε, τοποθετήσεις. Και ο Αρσένης, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς θέλουμε να συγχαρούμε τον οργανισμό για το έργο που κάνει. Υπάρχει ένα γεγονός που αναφέρεται στο διεθνή τύπο σχετικά με αυτούς τους ε, στα σκάφη και τους παρατηρητές και λέγεται ότι οι παρατηρητές μπορούν να καλέσουν μια επιθεώρηση στο πλοίο χωρίς όμως να μπορούν να καταγράψουν αυτές τις παρατυπίες που μπορεί να παρατηρήσουν. Ε, αυτό δεν είναι τεράστιο εμπόδιο στο έργο των επιθεωρητών, καθώς επηρεάζει την ε, ικανότητα τους να κάνουν ένα αποτελεσματικό έλεγχο. Επειδή πολύ συχνά τα αποδεικτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο φυσικά ε, δεν ε, τους δίνονται. Ίσως να γνωρίζετε ότι και ο Guardian έχει αναφέρει σε τέτοια περιστατικά. Ποια είναι η γνώμη σας από αυτού. Έχετε σκοπό να λάβετε κάποια δράση ή έχετε ήδη λάβετε δράση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκαρθία Πρεσέδο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη τόσο ενδελεχή παρουσίαση. Τρία συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτον, ένα σύντομο σχόλιο για τη συνεργασία του οργανισμού με άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Πρόσφατα, μία αντιπροσωπεία αλίας ε, του Κοινοβουλίου έχει πάει στην Ισλανδία. Ξέρετε, η Ισλανδία συνεργάζεται στον τομέα της παρακολούθησης στο πλαίσιο του Σέγγεν. Η δραστηριότητα στα πλαίσια Σέγγεν δεν έχει έχουν για κάποιες συμβατότητες με τις επιθεωρήσεις σε θέματα αλληλείας. Ρώτα λοιπόν, η Ισλανδία είναι μια χώρα υποψήφια για προσχώρηση. Δεν ε, θα ήταν σκόπιμο να συνεργαστεί μαζί μας και σε αυτόν τον τομέα. Δεν θα ήταν καλό να έχουμε ένα διαθρωμένο διάλογο και συνεργασία με αυτή τη χώρα. Δεύτερο ερώτημα για τις απορρίψεις. Αναφερθήκατε στις απορρίψεις χωρίς να μπείτε σε πολλές λεπτομέρειες. Ρωτώ, είναι δυνατόν να υπάρχει έλεγχος χωρίς δυσανάλογο ο κόστος σε ό,τι αφορά τις απορρίψεις πάντοτε. Και τρίτον, αναφερθήκατε σε ένα πιλωτικό project. Το πιλωτικό αυτό project είναι το ίδιο με αυτό που αναφέρεται, που, μάλλον που γνωρίζουμε ως εκστρατεία για τον τόνο στην Μεσόγειο, αναφέρεται σε κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Λομέν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά για αυτή την εντελεχή παρουσίαση που μας κάνατε. Θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό το έργο που κάνατε για τη βελτίωση της παρακολούθησης και εποπτείας Ευρωπαϊκής Ελίας και το συντονιστικό σας έργο και προσπάθεια είναι εξαιρετικές. Θα ήθελα ουσιαστικά να πω ότι Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ε, ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εφαρμοστούν τα μελλοντικά σας προγράμματα. Ε, να ρωτήσω λοιπόν κάτι για τον προπολογισμό του οργανισμού. Θεωρείτε ότι είναι αρκετός ο προπολογισμό για τα μελλοντικά σας σχέδια. Ιδίω αναφέρουμε στο κοινό σχέδιο ανάπτυξης ε, στην Μαύρη Θάλασσα και σε σχέση με την μελλοντική εφαρμογή του προγράμματος για την απαγόρευση των απορρίψεων. Να συμφωνήσω και με αυτά που είπε η κυρία Γκαρσία Ιέρο Καμπάγιο, ότι χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση του οργανισμού για τις επιθεωρήσεις που κάνει, όταν ε, μειώνει το προπολογισμό σχετικά με τη μίσθωση σκαφών, πώς μπορεί να γίνει αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Ρόντους συγγνώμη, δεν κατάλαβα το όνομά μου το ίδιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τόσο λεπτομερή παρουσίαση που μας κάνατε. Είπατε ότι τα αποτελέσματα του Συμβουλίου πριν από 14 ημέρες σαφώς αφορούν και την, τον δικό σας οργανισμό. Πώς βλέπετε τους ελέγχους μετά από αυτή την απόφαση. Επίσης, μιλήσατε λίγο για τις ε, δυνατότητες. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι τα κράτη αυτά που έχουν ακόμα δυνατότητες, πώς τις ε, καθορίζετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, θέλω να το ξέρω. Και επίσης, τα επιστημονικά στοιχεία που διαθέτεται είναι αρκετά, είναι επαρκή, είναι αξιόπιστα. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να υπάρχουν διαθέσιμα περισσότερα και πιο αξιόπιστα επιστημονικά στοιχεία εκεί που δεν αρκούν και δεν είναι καλής ποιότητας. Τελευταία ερώτηση. Θεωρείτε ότι σας αρκεί το προσωπικό, οι συνεργάτες που έχετε στη διάθεσή σας γιατί πραγματικά αυτό που όλοι θέλουμε είναι να χρησιμοποιούνται οι άνθρωποι και οι δυνατότητες που έχετε σαν οργανισμός με έναν τρόπο που να είναι πραγματικά αποτελεσματικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Σταυρό να απαντήσει εντάχει σε αυτές τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε και κύριοι. Στην κυρία Γκαρσία θα απαντήσω ότι τα κράτη-μέρη συνεισφέρουν όσον αφορά τα στοιχεία και τα δεδομένα βάσει των νομικών υποχρεώσεων που έχουν. Και βεβαίως το κοινό πρόγραμμα ειδικών επιθεωρήσεων και ελέγχων προϋποθέτει ότι αυτά τα στοιχεία και για τους ε, ελέγχους που γίνονται σήμερα και τους μελλοντικούς ελέγχους με ηλεκτρονικό τρόπο, αλλά και τους παρελθόντες ελέγχους, είναι απαραίτητο να είναι διαθέσιμοι και αξιόπιστα στοιχεία. Το πιλωτικό πρόγραμμα στο οποίο αναφέρθηκα, αναφέρεται στον τόνο, το κόκκινο τόνο και βεβαίως αυτό χρησιμοποιήθηκε γιατί είναι ενδιαφέρον σαν ε, βάση δεδομένων, περιορίζεται όμως στη Μεσόγειο σε αυτή την περίπτωση. Ο χώρος δηλαδή ήταν συγκεκριμένος και περιορισμένος. Ο συντονισμός ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικός, συντονισμός ε, του οργανισμού και με αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε πληροφορίες που κανονικά δεν χρησιμοποιούνται από τις αρχές ελέγχου της αλίας. Το αποτέλεσμα ήταν η βελτίωση αυτών των κοινών δυνατοτήτων που έχουμε για την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των ελέγχων και των επιθεωρήσεων. Βεβαίως, τηρούνται πάντα οι κανόνες προστασίας της ιδιωτικής ζωής και σας επαναλαμβάνω ότι ο απότερος σκοπός μας είναι πάντα η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων και η προστασία των αποθεμάτων. Τώρα, όσον αφορά τους παρατηρητές, υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τύποι παρατηρητών. Οι παρατηρητές Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του περιφερειακού ICAT έχουν δυνατότητα να αναφέρουν ανομαλίες παρατυπίες που εντοπίζουν ε, επιτόπου. Ο ρόλος ενός παρατηρητή περιγράφεται πλήρως στον κανονισμό των ελέγχων και των επιθεωρήσεων. Ο παρατηρητής λοιπόν, όπως καθορίζεται από τον κανονισμό του ICAT, αλλά και αυτό είναι θέμα, αν θέλετε, διαπραγμάτευσης στα πλαίσια του ICAT. Είναι ένας ρόλος που, αν θέλετε, ορίζεται πιο πολύ από τον ευρωπαϊκό κανονισμό παρά ότι από αυτά που προβλέπει ο ICAT. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Δεν μπορώ να μπω σε πολλές λεπτομέρειες για το θέμα αυτό. Τώρα, για τις απορρίψεις, απαντώ στον κύριο Σάντσες. Ο οργανισμός μπορεί να προτείνει κάποιες ε, σκέψεις και προτάσεις. Σήμερα χρησιμοποιούνται κάμερες εγκαταστημένες στα σκάφη και μπορεί κανείς να διασταυρώσει τα στοιχεία, δηλαδή επιπλέον από τις πληροφορίες που έχουμε από τις κάμερες, να χρησιμοποιήσουμε κάποια σκάφη μοντέλα Βάσει των στοιχείων λοιπόν αυτών των σκαφών, της δραστηριότητας αυτών των σκαφών, ορίζονται κάποιες ποσότητες, κάποια ποσοστά και βάσει αυτών των υπολογισμών θεσπίζονται και οι ποσότητες των απορρίψεων, τα ποσοστά των απορρίψεων. Άλλη ερώτηση. Συνεργασία με άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα. Συνεργαζόμαστε με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας των Θαλασσών και την Frontex. Με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας και τον ειδικό Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Μεσόγειο. Συνεργαζόμαστε για τον τόνο της Μεσογείου και ειδικότερα, όπως σας είπα με πολλές λεπτομέρειες στην παρουσίασή μου, έχουμε μια εξαιρετικά οργανωμένη συνεργασία. Για την Frontex χρησιμοποιούμε πολλές φορές εξοπλισμό, όπως σας ανέφερα την περίπτωση ενός ναυλωμένου σκάφους, το οποίο μας διαθέτει η Frontex. Κατά τα άλλα δεν έχουμε συνεργασία οργανωμένη θεσμοθετημένη με άλλους οργανισμούς. Ε, το σκάφος το οποίο έχουμε να ναυλώσει και χρησιμοποιούμε είχε σημαία Ισλανδική. Πρόκειται για μια τεχνική συνεργασία, αποτελεσματική και αν κάποια στιγμή στο μέλλον εξελιχθούν οι σχέσεις μεταξύ Ισλανδίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, βεβαίως και είμαστε ε, διατεθειμένοι να συνεργαστούμε και με την Ισλανδία και με άλλες τρίτες χώρες. Προϋπολογισμός. Το 2011 αναλώθηκε 90% του προϋπολογισμού των διαθέσιμων πόρων και σήμερα αντιμετωπίζουμε κάποιες επιπλέον δυσκολίες γιατί ο οργανισμός όπως ξέρετε, έχει μάλλον πνευματική δραστηριότητα και οι περικοπές σαφώς και θα έχουν άμεσες επιπτώσεις σε αυτή τη δραστηριότητα. Αν αναγκαστούμε να αναπτύξουμε συστήματα πληροφοριών για τα κράτη-μέλη, καταλαβαίνετε ότι ο προϋπολογισμός θα πρέπει να αυξηθεί σημαντικά κατά κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Το θέμα των ε, δυνατοτήτων και των πλεονασμάτων αυτό είναι κάτι που βεβαίως δεν μπορεί να μετρηθεί μόνο σε σχέση με το τονάζ και τις δυνατότητες του στόλου. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι υψηλός 27 χρόνια. Υπάρχει όμως και το θέμα της σύγχρονης ή απαρχαιωμένης τεχνολογίας που χρησιμοποιούν τα σκάφη αυτά. Υπάρχουν εκθέσεις για το θέμα αυτό και είναι δύσκολο κανείς να πάρει μια συγκεκριμένη θέση. Συμφωνώ όμως ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Τα επιστημονικά δεδομένα για τα κοινά σχέδια, κοινά προγράμματα, τα στοιχεία που διαθέτουμε είναι εξαιρετικά αξιόπιστα παραδείγματο χάρη για την προετοιμασία του κοινού προγράμματος για το Σολομό. Διαθέτουμε εξαιρετικά αξιόπιστα επιστημονικά στοιχεία. Όπως ξέρετε θα υπάρξει το 2012 αναθεώρηση από την Επιστημονική Επιτροπή το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο της επιστημονικής δραστηριότητας και αναθεώρηση της ε, διαχείρισης από το ΆΙΚΑ για τον κόκκινο τόνο. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι τα κράτη-μέλη στηρίζουν και συνεισφέρουν στη δραστηριότητα του οργανισμού μας με πολύ θετικό και αλληλέγγυο τρόπο και νομίζω ότι εκτιμούν τον συντονιστικό ρόλο του οργανισμού. Όσον αφορά την περιφερειακή προσέγγιση, σαφώς και θα πρέπει να βρούμε και άλλες δραστηριότητες οι οποίες να συμπεριληφθούν ε, και αυτό οπωσδήποτε θα έχει και δημοσιονομικές επιπτώσεις ε, για τον οργανισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σεωχέ. να σας αποχαιρετήσουμε και θα τα ξαναπούμε τον επόμενο Οκτώβριο. Λοιπόν, συνεχίζουμε άμεσα στις ηλεκτρονικές ψηφοφορίε, καθώς έχουμε ένα μακροσκελή κατάλογο. Παρακαλώ να έχετε έτοιμη την κάρτα σας και πάντοτε απόλυτη προσοχή ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ταχύτατα. Πρώτα απ' όλα ξεκινούμε με το σημείο 5 πολιτέ σχέδιο για το απόθεμα Σολομού της Παλτικής και την αλληλευτική εκμετάλλευση του συγκεκριμένου αποθέματος. Είμαστε έτοιμοι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Τροπολογία υπαριθμών 7. Αρχή ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Τροπολογία 6. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία NV 12. Αρχή. ΕΝΒΙ 12. Ψηφίζουμε. Κύριε Κούν. Η 43 έχετε αποσυρθεί. Ναι, ναι, λέει ο Πρόεδρος. Ε, Εμφανίζω τον κατάλογο ως ε, ότι έχει αποσυρθεί. Γι' αυτό δεν την ανέφερα. Λοιπόν, ψηφίζουμε την ένδυ 12. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Είναι 12 υπέρ και 12 κατά. Τροπολογία 8 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 1, αρχή ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 2, ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβασμός 3. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 50. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 51. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 52. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 12. Ψηφίζουμε. Τροπολογία 12. Πέρας. Εγκρίνεται. NV16. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. NV17. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 54. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 13. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. ΕΝΒΙ 18 Α, με συγχωρείτε, εγκρίθηκε η Πάμε στον συμβασμό 4 κατευθείαν. Ψηφίζουμε. Πέρας. ΕΝΒΙ NV21. Πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Όχι λοιπόν, τροπολογία 56. 56 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 57. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 1. Ψηφίζουμε. Είναι σαν συμβασμός. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Ψηφίζουμε. 16, συγγνώμη, τροπολογία 16 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. NV22 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 59 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. NV23 Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 60, συν προφορική 3 σε 2 τμήματα. Πρώτο τμήμα, ψηφίζουμε. Πέρας. Εκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 62. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 61. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. NV25. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. NV24 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 65 ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε την 65. Πέρας. Εγκρίνεται. 64. Όχι, καταπίπτει. 63. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 66. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 67 ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα, το πρώτο τμήμα της 67, πέρας, εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα, πέρας, απορρίπτεται. 68. Πέρας. Εγκρίνεται. ΕΝΒΙ Εγκρίνεται. NV27. NV27 επαναλαμβάνει ΕΝΒΙ 27. Ψηφίσαμε την NV26 που εγκρίθηκε και είμαστε στην NV27 άρθρο 16. Εκτός μικροφώνου η ανταλλαγή απόψεων. NV λοιπόν 27 κατά άρθρο 16. Ψηφίζουμε. nv λοιπον 27 το αρθρο Εγκρίνεται. 70 λέει ο πρόεδρος. 72. Λάθος. 72. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Ένδυ 29. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 75. Πέρας. Εγκρίνεται. 76. Πέρας. Εγκρίνεται. 77. Πέρας. Εγκρίνεται. NV30 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 20. Πέρας. Απορρίπτεται. 78. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 80. Πέρας. Εγκρίνεται. 21. Πέρας. Εγκρίνεται. NV31. Πέρας. Εγκρίνεται. 82. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 22. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 83. Πέρας. Εγκρίνεται. 23. Πέρας. Εγκρίνεται. 24. Πέρας. Εγκρίνεται. 25. Πέρας. Απορρίπτεται. 84. Πέρας. Απορρίπτεται. 85. Πέρας. Απορρίπτεται. Όχι, όχι, λάθος. Ούτως ή άλλως απορρίπτεται. 86. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στα παραρτήματα. NV33. Πέρας. Απορρίπτεται. Εκτιμώντας. NV1. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. NV2 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Πέρας. Απορρίπτεται. 28. Εκτός μικροφώνου. Οι στοιχομηθίες να το επαναλάβουμε. NV2, δεύτερο τμήμα. Επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία. Εντάξει. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 28. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 27. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 29. Πέρας. Εγκρίνεται. 30. Πέρας. Απορρίπτεται. NV4. Όχι, με συγχωρείτε. NV5. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 32 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 35. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. NV6 πέρας εγκρίνεται 36 πέρας εγκρίνεται προφορική 2 Κρίστενσεν ψηφίζουμε πέρας εγκρίνεται NV8 πέρας εγκρίνεται 40 ψηφίζουμε πέρας εγκρίνεται 41 πέρας Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε την ομοθετική πρόταξη όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται ομοφόνος και το ψήφισμα στο σύνολό του. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Θερμά συγχαρητήρια στον εισηγητή. Περνάμε στο επόμενο σημείο μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής θεμελιώδης ανακοίνωση. Έκθεση του κύριου Σαλαβράκου. Με πολλές τροπολογίες και εδώ. Θα είμαστε εξίσου προσεκτικοί όπως και με την πρώτη. Να ξεκινήσουμε την τροπολογία 40. Α, μισό λεπτό, ναι, μάλιστα, παρακαλώ. Επειδή το μηχανήμα μου έχει κάποιο πρόβλημα, στην προηγούμενη ψηφοφορία ενώ χτύπησα πράσινο, πήγε κόκκινο. Είναι ομοφωνία επομένως, Το ένα που παρουσιάστηκε σαν κόκκινο ήταν εκλάθος του μηχανήματος στην προηγούμενη ψηφοφορία. Είναι ομοφωνία. Ναι. En Πάντω, αν συνεχίσει να μην λειτουργεί σωστά το μηχάνημά σα, καλό θα ήταν ίσω να αλλάξετε θέση για να αποφύγουμε αυτό το πρόβλημα. Ωραία, έτσι αποφεύγουμε να ξανασυμβεί αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σαλαβά και ξεκινάμε λοιπόν. Ψηφίζουμε την έκθεσή σας. Τροπολογία 40. Έναρξη ψηφοφορίας. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 41. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 42. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 43. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. τροπολογία 44 και 45 ταυτόσιμες άναξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνονται. Τροπολογία Ρέτζι 1. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Όχι, πηγαίνουμε στην 46 τροπολογία τώρα. Πέρας ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 48. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Να ξαναρχίσουμε με τη 48. 48 έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 52. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβεβαστική 6. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Πού πηγαίνουμε τώρα. 57. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 61. Υπέ, άρχεται η ψηφοφορία, συγγνώμη. Πέρας. Απορρίπτεται τροπολογία Ρέτζι 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογίες 64, Rage 22, ταυτόσημες. άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτονται. Συμβιβαστική 8. Με μία προφορική τροπολογία. Την έχετε. Παρακαλώ. Χωρίς μικρόφωνο. Δεν δέχομαι την προφορική τροπολογία. Πρόεδρος, μάλιστα. Συμβιβαστική λοιπόν 8 ως έχει. Άρχεται τη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 66. Άρχεται τη ψηφοφορία. Πέρας. Όχι, εντάξει, περιμένουμε. Λοιπόν, 66. 66. Τροπολογία 66. Τι πρόβλημα υπάρχει. Ψηφίσατε όλοι. ψηφοφορία σου. Απορρίπτεται. Τροπολογία 68. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 71 με 72 ταυτόσιμες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτονται. Τροπολογία 73. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 75. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 77. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 78. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 80. Άρχεται η ψηφοφορία. 80. Πέρας. Απορρίπτεται. 83. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 84. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 86. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Πού πάμε. 90. Όχι. Ούτε εκεί. 91. 91. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 92. 93. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 101. 101. Άρχεται ψηφοφορία. Το βρήκατε, εντάξει. Λοιπόν, πέρασε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12. Άρχεται ψηφοφορία. Παρακαλώ κυρία Λέβιν, θέλει κάτι. θα μπορούσε να ψηφιστεί ως προσθήκη σε συμβαστική 11, η τροπολογία 108. Όχι, λέει αν η συμβιβαστική εγκριθεί, καταπίπτει. Βέβαια λέει εδώ ότι μπορεί να ψηφιστεί ως προσθήκη. Να ψηφίσουμε δεν ξέρω. Λοιπόν, από ότι μου εξηγούν. Από ό,τι φαίνεται θα μπορούσε να ψηφιστεί ως προσθήκη, αλλά ως προσθήκη στις τροπολογίες, εφόσον δεν είχε εγκριθεί η συμβιβαστική 11. Αφού εγκρίθηκε η συμβιβαστική 11, καταπίπτουν οι άλλες, άρα δεν μπορεί να προσθεθεί σε αυτές οι 108. Καταλάβατε τι είπα. Λοιπόν, τι κάναμε, ψηφίσαμε. Ψηφίσαμε τη 12. Όχι, αρχίζουμε πάλι την ψηφοφορία επί της ε, συμβιβαστικής 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 120. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 121. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 124. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 123. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 125. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 126. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 127. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 128. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 131. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 134. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 135. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 136. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 137. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 139. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολόγια 140. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 141. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική υπερθών 14 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτό το πρώτο. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτό και το δεύτερο. Είμαστε τώρα στην τροπολογία 145. Άρχεται η ψηφοφορία. 145. Πέρας. «145. Κρατάω λίγο ακόμη ανοιχτή την ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Να επαναλάβουμε. Λοιπόν, έναρξη της ψηφοφορίας για την 145. Πέρας. Απορρίπτεται. 146. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. 147. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 148. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 149. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 150. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παρακαλώ. Κυρία Λάβιν. Ε, δεν έχει και τόσο σημασία, απλά δεν ψήφισα. Ευχαριστώ. 151 ε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. 154 Χάγκλουντ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 155 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 157. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 160. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 161. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 165. 165. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 166. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17. 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και περνούμε στην τροπολογία 178. 178. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 180. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 182. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία ΔΕΒΕ 7. Άρχεται η ψηφοφορία. ΔΕΒΕ 7. Παράγραφος 22F. Η ΣΥΓΜΑΤΑΦ. Έχουμε δύο από την ΤΕΒΕ, την 7 και την 8. Κατάξει, τα βρήκατε. Λοιπόν, ψηφίζουμε την ΤΕΒΕ 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. ΤΕΒΕ 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογίες 184-185 ταυτόσιμες άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτονται. Δεν λειτουργεί, το μηχάνημά μου, λέει. Λοιπόν, συμβιβαστική 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 191. 1, 9, 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 195. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 196. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 197. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 198. Όχι, όχι. Συγγνώμη. 199, 200, 201, 202 Ούτε και αυτές, μάλιστα. Πού πάμε λοιπόν. Πάμε, πάμε. Ναι, κύριε Αρσένη. Εκτός μικροφώνου. Κύριος Αρσένης. Ήθελα στην προηγούμενη ψηφοφορία να ψηφίσω κατά, αλλά ήταν αδύνατο να ψηφίσω. Δεν, δεν μπορούσα να... δεν λειτουργούσε. Δυστυχώ, ο πρόεδρο, τώρα δεν μπορούμε να επαναλάβουμε την ψηφοφορία, τέλο πάντων. Λοιπόν, πηγαίνουμε στη 207 τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 19. Συμβιβαστική 19 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία ΔΕΒΕ 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 211. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 212. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 213. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 214. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 215. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 216. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 217. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 218. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 219. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 220. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 221. 221. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 222. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται, εγκρίνεται, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 223. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 229 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 230 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 231 άρχεται. Πέρας εγκρίνεται. 232 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 233 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 234 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 235 της ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 236 της ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 237 της ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 238 άρχεται. Λύνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 239 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 240 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 241 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 242 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 243 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 245. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 246. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 247. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 248. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 249. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 250. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 251. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 252, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 253, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 21, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Τώρα, περνάμε στην τροπολογία Χάγκλουντ υπαριθμών 262. 262. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 263. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 264 άρχεται ψηφοφορία. Α, συγγνώμη, έχει κρίνει. Λοιπόν, 264 τελικά. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 265 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 266 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 267 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 268 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 269 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 270 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 271. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 272 τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 273. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 274. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 275. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 276. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 277 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 278 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ρέτζι 19 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ρέτζι 20 άρχεται. Πέρας εγκρίνεται. Τροπολογία 279, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 280, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 281, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 282 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 283 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 284 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 285 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 286. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεύε 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύε 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ντεβε 12, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ντεβε 13, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ντεβε 14, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 23 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 27. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4 συμβιβαστική. Συμβιβαστική 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Τροπολογία 33. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 34. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 35. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 36. Άρχεται. Πέρας. εγκρίνεται. 37. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 38. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 39. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 21 ψήφοι υπέρ, 2 κατά, 2 αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Σαλαβράκου. Περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία για το διάμεση έκθεση ενώ ψηθεντή η έκταση στη διαδικασία έγκριση πολιτού σε δημοσιονομικού πλαισίου, εισηγητή ο κύριο Φερέιρα. Εδώ έχουμε λίγε τροπολογίε. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση, να ξεκινήσουμε αμέσω. Τροπολογία 1. Ψηφίζουμε. Έκθεση γνωμοδότηση συγγνώμη, Φερέιρα. Τροπολογία 1. Πέρα ψηφοφορία εγκρίνεται. Δύο ψηφίζουμε σε δύο τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Πέρας. Εγκρίνεται επίσης. Τροπολογία 4 ψηφίζουμε. Πέρας. Εκρίνεται. Τροπολογία 5 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 7 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 9. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 10. Πέρας. Εγκρίνεται. 11. Πέρας. Εγκρίνεται. 12. Πέρας. Εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε τώρα την γνωμοδότηση όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ομοφόνος. Συγχαρητήρια κύριε Φερέιρα. Τέλος η ψηφοφορία λέει ο Πρόεδρος. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, το σημείο 17, όπως ήδη είχαμε ανακοινώσει. Έκθεση Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεκτικό των πολιτικών ανάπτυξης. Ah, perdón, perdón, perdón. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος. Έχουμε και, άλλες, άλλη ψηφοφορία να κάνουμε. Perdón, ha sido un error mío. Λάθος σφάλμα δικό μου. Έχουμε τη συμφωνία του Τριλόγου 20 Ιουνίου για τα μέτρα κάτω χωρών που επιτρέπουν τη εξαγωγή μη βιώσιμης αελίας με στόχο τη διατήρηση των ηχθοποθεμάτων. Η συγκρίτηση ο κύριος Γκάλαγκερ. Ψηφίζουμε εν λόγω. Έχετε μπροστά σας την πρόταση, οπότε θέτουμε σε ψηφοφορία ε, το συμβιβασμό. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται ομοφόνος. Συγχαρητήρια κύριε και δεν ήταν και εύκολο αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, τώρα ναι, τώρα περνάμε στο σημείο 17, όπως ήδη ανακοίνωσα πριν. Η συγγητής ο κύριος Φερέιρα θα μας παρουσιάσετε λοιπόν κύριε Φεραίρη το σχέδιο γνωμοδότησης που εκπονήσατε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Καλά. Ας φύγουν όσοι δεν επιθυμούν να ακούσουν για να έχουμε ισχύα. Κύριε Φερέιρα, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομο. Ήδη είχαμε την ευκαιρία για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για αυτή την γνωμοδότηση που αφορά τη συνοχή της αναπτυξιακή πολιτικής ε, πρόκειται για έναν τομέα ε, στον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να προσεγγίσει οριζόντια, δηλαδή με μία δέσμη, ε, με ένα πλέγμα πολιτικών. Θα κάνω κάποια γενικά σχόλια για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Ουσιαστικά, θεωρούμε ότι είναι πολύ περιορισμένη η προσοχή που δίνεται σε αυτό το θέμα, μάλιστα στην τελευταία συνεδρίαση είχαμε συζητήσει και την έκθεση της ίδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έκθεση αξιολόγησης συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις πολιτικές ανάπτυξη. Ε, δίνει τόσο μεγάλη σημασία σε αυτή την έκθεση που δεν τη μεταφράζει καν σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Αν δεν κάνω λάθος, φοβούμαι, αλλά μόνο στα αγγλικά μπορεί να το βρει κανείς. Να, ένα πρώτο αρνητικό σημάδι. Σε ό,τι αφορά την αλληλεία, η συνοχή των πολιτικών ανάπτυξης μπορούν να συνοψιστούν σε τρεις άξονες σε ό,τι αφορά την αλληλεία πάντοτε. Πρώτα απ' όλα, βιωσιμότητα των αποθεμάτων και ο αντίκτυπος των αλληλευτικών δραστηριοτήτων στις αλληλευτικές κοινότητες στις υποανάπτυξη χώρες. Δεύτερος άξονας είναι οι συμφωνίες συνεργασίας στην αλληλευτική πολιτική με τις χώρες και οι οικονομικές αποζημιώσεις προς αυτές τις χώρες και τρίτη πτυχή άξονας είναι η εναρμόνιση στα πλαίσια ενός περιφερειακού συστήματος ε, βιώσιμης διαχείρισης ε, των αλληλευτικών πόρων. Στην ε, γνωμοδότηση που έχετε μπροστά σας για διαφόρους περιορισμούς που είχαμε σε αυτή τη φάση, βλέπετε ότι αναφερόμαστε μόνο στα θέματα των συμφωνιών συνεργασίας θέματα αλληλείας. Περίπου το ίμιση των στόλων που αλλιεύουν ε, στη, στα διεθνή ύδατα διέπονται από αυτές τις ε, ε, συμφωνίες, διμερείς συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες αλλιές. Θέλω να επισημάνω και ενώπιση των τροπολογιών που θα υποβληθούν, σε όλο αυτό το τομέα της αλίας που κινούνται εκτός των συμφωνιών αυτών, είναι θέματα τα οποία θα τα αναφέρω στη γνωμοδότησή μου. Ε, δεδομένου των διαφόρων περιορισμών, εγώ ε, εστίασα στις διάφορες συμφωνίες αλίας, αναφέροντας ότι λυπόμεθα ιδιαίτερα για τις ελλείψεις και τα κενά που υπάρχουν σε επιστημονικό και τεχνικό επίπεδο στο λεγόμενο ε, τομέα της ε, τομεακής στήριξης, ιδίως ό,τι αφορά τη στήριξη της αναπτυσσόμενης χώρες. Αυτό βεβαίω μεταφράζεται ουσιαστικά στη μεταφορά ε, κονδυλίων, ε, ενισχύσεων, στήριξη προ αυτέ τι χώρες. Βεβαίω, αυτό που ισχύει σήμερα είναι μια πολύ αυστηρή ανάγνωση ερμηνεία των συμφωνιών αυτών. Οι συμφωνίε αυτέ έχουν ουσιαστικό στόχο την υποστήριξη του αλληλευτικού τομέα ε, σε αυτέ τι χώρε. Γι' αυτό και γι' αυτό ονομάζονται και τομεακέ συμφωνίε ουσιαστικά. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια δέσμη μέτρων και δράσεων ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε καλύτερα σε πνεύμα συνεργασίας αυτά τα σύμφωνα με χώρες. Αυτό ε, βεβαίω θα πρέπει να προβλέπει και μηχανισμό διορθωτικό, δηλαδή να υιοθετούνται και διορθωτικά μέτρα όταν εντοπίζονται προβλήματα γιατί πολλέ φορέ υπάρχει απόκληση ανάμεσα στι συμφωνίε και την πρακτική του εφαρμογή. Εδώ χρειάζεται συνεργασία της χώρε. Βεβαίω. χρειαζόμαστε πάντοτε επικυροποιημένα επιστημονικά στοιχεία και για τα αποθέματα και για τη συνολική αλληλευτική προσπάθεια στα ύδατα κάθε χώρα. Είναι ένα θέμα που τίθεται συνεχώς στο τραπέζι των συζητήσεων. Το θέμα της ε, παράνομης, λαθρέας και άναρχης ε, αλίας και τέλος μια καλύτερη διάρθρωση αυτών των συμφωνιών συνεργασίας στο τομέα Ελίας σε σχέση, σε ακολουθία με άλλες αντίστοιχες συμφωνίες συνεργασίας σε άλλες τομιακές πολιτικές. Αυτά ουσιαστικά είναι τα μείζωνα σημεία της Απλά θέλω να επισημάνω και πάλι ότι κάποια στοιχεία που δεν αναφέρονται αυτή τη στιγμή στην ομοδότηση και χρήζουν εξέταση, ιδίω ότι αφορά την ελευθερική δραστηριότητα εκτό των συμφωνίων συνεργασία που είναι πάνω από το ίμιση της αλίας που γίνεται εκτός ενωσιακών υδάτων και γίνεται σε ύδατα υποανάπτυξη χωρών, έω τώρα δεν είναι θέματα που έχουν συμπεριληφθεί στη γνωμοδότηση για διαφόρους ε, λόγους, αλλά θα επιληθεί αυτό το ζήτημα με την υποβολή τροπολογιών και τη συζήτησή τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φερέρα. η κυρία Λεβέν. Ε, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Φερέρα για την εξαιρετική αυτή παρουσίαση της γνωμοδότησής του. Εγώ παρακολουθώ το θέμα από την Επιτροπή Ανάπτυξης και στηρίζω σε μεγάλο βαθμό τις προτάσεις του εισηγητή. Θα κάνουμε κάποιες τροπολογίες. Ένα θέμα που μου φαίνεται πολύ σημαντικό ομιλούμε για τις αναπτυσσόμενες χώρες, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι πραγματικά εξυπηρετείται εδώ ο σκοπός ε, τον οποίο έχουμε θέσει. Δηλαδή ότι στηρίζεται η αλληλευτική πολιτική στην χώρα τους και ότι τα κονδύλια αυτά δεν ε, τροφοδοτούν ε, άλλα, άλλες δραστηριότητες, διαφθορά κτλ. Το θέμα λοιπόν της διαφάνειας είναι πολύ σημαντικό καθώς και το θέμα της εμπλοκής, της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών αυτών των χωρών, των αναπτυσσόμενων χωρών, οι οποίοι θα πρέπει να είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Οι διαπραγματεύσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα θα πρέπει να είναι διαφανείς, Να υπάρχει δηλαδή πρόσβαση στα στοιχεία των διαπραγματεύσεων, στις εντολές κτλ. Και γνωρίζουμε ότι στις ε, τρίτες χώρες, στις αναπτυσσόμενες χώρες, πολλές φορές δεν υπάρχει ενημέρωση. Ακόμα και το κοινοβούλιο πολλές φορές ε, δεν έχει ε, καμία συμμετοχή στην διαπραγμάτευση και στην όλη διαδικασία. Ξέρουμε λοιπόν ότι και από άλλους τομείς όπως το τομέα της εξορρυκτικής βιομηχανίας είτε την υλοτομία, τα δάση, ότι πραγματικά δεν υπάρχει συμμετοχή της κοινωνίας και των δημοκρατικών θεσμών στις ε, χώρες αυτές όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις. Όσον αφορά λοιπόν την εξωτερική διάσταση της αλληλευτικής πολιτικής και την μεταρρύθμιση, θα πρέπει να υπάρξει, αν θέλετε, μια διαφορετική αντιμετώπιση της συμφωνίας σε σχέση με το κομμάτι το επιχειρηματικό. Και μόνο αν ε, ξεκαθαρίσουμε, αν θέλετε, αυτήν την οικονομική πτυχή και δεν μπορούμε να λέμε αν θέλετε, με τόσο ξεκάθαρο τρόπο ότι η αναπτυξιακή βοήθεια που θα τους παρέχουμε εξαρτάται από την δυνατότητα που μας δίνουν να έχουμε πρόσβαση στα δάση τους ή ε, τους φυσικούς τους πόρους, την αλία κτλ. Δεν είναι δυνατόν. Θα πρέπει πραγματικά τα δύο αυτά θέματα να είναι ξεχωριστά και δεν μπορούμε, είναι θέμα αρχής, δεν μπορούμε να το θέτουμε σαν προϋπόθεση ότι θα δοθεί δηλαδή αναπτυξιακή βοήθεια μόνο και εφόσον έχουμε πρόσβαση στους φυσικούς τους πόρους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλες τις διαπραγματεύσεις με τις τρίτες χώρες, όχι μόνο με τις αλλιευτικές συμφωνίες. Θα πρέπει να υπάρχει μια οικονομική συμφωνία που να καλύπτει το θέμα της αλληλείας. Και είναι πολύ σημαντικό οι ίδιοι οι πλειοκτήτες να χρηματοδοτούν σωστά και να μην τροφοδοτεί, να μην χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση την ε, οικονομική αυτή διάσταση της δραστηριότητας. Αλλιώς βλέπουμε ότι οι τρίτες χώρες δεν ε, εποφελούνται όσο θα έπρεπε από αυτές τις επιδοτήσεις. Θα πρέπει λοιπόν εδώ πολλά βήματα να γίνουν η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει σαφώς να βελτιώσει όλες αυτές τις συμφωνίες αναπτυξικής βοήθειας και αλληλευτικής πολιτικής. Και εδώ το άρθρο 208 της συνθήκης προβλέπει ότι όλες οι κοινοτικές πολιτικές που έχουν επιπτώσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι αντικρουόμενες πολιτικές σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί στην αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική αρχή και χαίρομαι διότι αυτό ακριβώς κάνει και πρεσβεύει και ο εισηγητής. Επαναλαμβάνω λοιπόν, θα υποβάλουμε τροπολογίες για αυτή την εξαιρετική γνωμοδότηση και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτή τη γνωμοδότηση. Ξέρετε, στα πλαίσια τόσων γνωτήσεων και τροπολογιών που έχουν υποβληθεί το τελευταίο διάστημα, ε, σαφέ σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προωθεί και υποστηρίζει την βιωσιμότητα Αναλύοντας τον αντίκτυπο που έχουν αυτές οι συμφωνίες ε, στις αλληλευτικές κοινότητες, εγώ θέλω να επισημάνω ότι όταν μιλούμε για αντίκτυπο, επειδή δίνεται μια αρνητική χρειά στην γνωμοδοτησία του. Ο αντίκτυπο δεν είναι πάντα αρνητικό. Υπάρχουν κάποιε συμφωνίε αλλίε με τι χώρε που έχουν και θετικέ συνέπειε, θετικό αντίκτυπο. Πιστεύω ότι ε, ναι, μεν εγώ συμφωνώ ότι είναι καλό που αναλύεται τις ε, συνέπειες αυτών των συμφωνιών σε αλληλευτικές αυτές ε, κοινότητες. Καλό είναι οι συνέπειες που θα αναλύσουν να είναι και θετικέ και αρνητικέ. Σε ό,τι φορά τι εφιστάμενε συμφωνίε με αυτές τις τρεις χώρε, θεωρούμε ότι η ίδια κοινότητα πολιτών θα πρέπει να αντιδράσει και να ζητήσει δύο είδου συμφωνίε. Είναι σημαντικό να υπάρχει ε, ακολουθή και συνεκτικότητα με τη συμφωνία σύνδεσης, διότι έχει καταστεί ε, σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις διάφορες συμφωνίες με τρίτες χώρες δεν ακολουθεί μία συνεκτική πολιτική σε θέματα ανάπτυξη με τις τρίτες χώρε. Θέλω λοιπόν και όσο σημαντικό να υπάρχει ενημέρωση, να υπάρχει διαφάνεια στα δεδομένα, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εντοπίσουμε τα καλά και τα κακά ε, στις πολιτικές μας για να μπορέσουμε να προτείνουμε και καλύτερες λύσεις στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά κάποια επιμέρους σημεία της οτομοδότησης που αναφέρονται ιδίω στην παράνομη αλία, πιστεύω ότι χρειάζεται και σε αυτή η γνωμοδότηση κάτι αντίστοιχο με αυτό που πριν για τον αντίκτυπο. Όταν μιλάμε για παράνομη αλία, ε, θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση, πιστεύω, πού και ποιοι κάνουν αυτή τη δραστηριότητα. Ποια σκάφη, ποια λευτικά σκάφη κάνουν σε μεγάλο ποσοστό αυτή την παρανομία Η ίδια η Κομισιόν σαν αναλύει πάντοτε ακριβώς πού έγκαιται το ζήτημα της παρανομίας και αυτό δεν αφορά κατά κύριο λόγο τα ευρωπαϊκά αλληλευτικά σκάφη. Θεωρώ λοιπόν στην παράγραφο 6 του κειμένου σας, όπου αναφέρεστε στην αλία Αγίου την παράνομη λαθρέα και άναρχη Ναι, συμφωνώ ότι ένα φαινόμενο πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αλλά καλό είναι να κάνετε μια κάποια μνήμα στις πρακτικές ε, των ε, ευρωπαϊκών αλληλευτικών στόλων. Για τροπολογίες τώρα. σχετικά με την εξωτερική διάσταση, να εμεί θέλουμε κάποιε τροπολογίε ώστε να υπάρχει μια καλύτερη ακολουθία στο κείμενό σα. Διότι υπάρχουν ποιε δηλώσει των εφοπλιστών, και αναφέρομαι στα σχόλια τη κυρία Λόβερ. διότι οι εφοπλιστές δείχνουν έτοιμοι να δώσουν πιο πολλά χρήματα σε αυτές, για την εφαρμογή αυτών των συμφωνιών Άρα υπάρχει μια θετική στάση και από το κλάδο και από την πλευρά των πλειοκτητών. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει μια θετική αντιμετώπιση. Θα υποβάλουμε λοιπόν κάποιες τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Σημαντικό είναι να υπάρχει, να υπάρχει περισσότερος και αποτελεσματικότερος έλεγχος και καλό είναι να αναλύουμε τις συνέπειες και τι θετικέ και τι αρνητικέ. Αν ζητούμε εμεί συνεκτικότητα και ακολουθεί από του άλλου, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δώσουμε εμεί το καλό παράδειγμα. Συνεχώ εμεί διαπιστώνουμε ότι οι άλλοι δεν ακολουθούν, α, ε, ε, ακολουθεί, δεν ακολουθούν ακολουθεί και συνεχτική πολιτική. Ε, α το κάνουμε εμεί πρώτα απ' όλα. Καλύτερα να προτείνουμε λύσει στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Με αυτόν τον τρόπο θα κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν επιθυμεί να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική αρχή, έννοια, που βεβαίως περιέχει η συνθήκη και είναι πάρα πολύ σημαντικό να την ακολουθήσουμε στην αλληλευτική πολιτική. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ευθύνες η Ένωση για να υπάρξει μια τέτοιου είδους ε, αλλιευτική πολιτική και εκτός των χωρικών ε, υδάτων της ε, κοινότητας. Γι' αυτό και μιλούμε για την εξωτερική διάσταση της αλλιευτικής πολιτικής και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα για τις προτάσεις του κυρίου Φερέιρα, τον οποίο ευχαριστώ, Είπατε ότι οι συμφωνίες ουσιαστικά σημαίνουν μεταφορά κονδύλιων. Ε, διαφωνούμε με αυτή την ε, άποψη του εισηγητή. Από το 2004 δεν υπάρχουν ε, καθαρά εμπορικές συμφωνίες. Σήμερα μιλάμε για εταιρική σχέση. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική πτυχή των συμφωνιών μας. Αυτή η εταιρική σχέση έχει σαν σκοπό να αναπτύξει αυτή την αλληλευτική πολιτική, την καλύτερη διακυβέρνηση, ιδιαίτερα με τις χώρες αυτές με τις οποίες έχουμε συνάψει αλληλευτικές συμφωνίες. 30% της χρηματοδότησης αυτών των αλληλευτικών συμφωνιών ουσιαστικά κατευθύνεται και τροφοδοτεί την στήριξη αυτού του τομέα. Στις διάφορες λοιπόν χώρες με τις οποίες συνάπτουμε συμφωνίες χρηματοδοτούμε την ανάπτυξη επιστημονικής έρευνας, διαχείριση των αλλιευμάτων, έλεγχος και επιθεώρηση, υποδομές, διοικητική υποστήριξη και υγειονομική, υγειονομικός έλεγχος. Δεν θα σας δώσω όλο τον κατάλογο των επιτυχημένων εταιρικών σχέσεων, αλλά πιο συγκεκριμένα για το μηχανισμό Όσον αφορά το VMS παραδείγματο χάρη, ξέρετε ότι οι αλήθειες έχουν γίνει πολύ πιο αποτελεσματικοί χάρη στη χρηματοδότηση και στους εξοπλισμούς αυτούς. Επίσης, όσον αφορά τα πληρώματα και την χρησιμοποίηση του εγχώριου πληθυσμού. Αυτό είναι κάτι που βοηθάει πάρα πολύ στην ανάπτυξη των τρίτων χωρών. Η ανάπτυξη των φυσικών πόρων και η εξαγωγή των φυσικών πόρων αυτών των χωρών. Κάτι που βεβαίως δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του το επίπεδο ανάπτυξης των χωρών με μεγάλες διαφορές. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας και όλες τις άλλες προτεραιότητες αναπτυξιακές οι οποίες πολλές φορές βρίσκονται σε άλλους τομείς και όχι στην αλία. Δεν είναι εύκολο να αναπτύξει κανείς ε, επίσης ε, έναν στόλο, εραστητεχνικό ή μη τεχνικό, επίσης δυνατότητες διατήρησης, ε, αποθήκευσης και κατάψυξης. Μιλήσαμε για διαφάνεια, για πρόσβαση στα δεδομένα. Η αξιολόγηση είναι πάρα πολύ σημαντική και πρόκειται για μια προϋπόθεση για την ε, ανανέωση των συμφωνιών. Προσπαθούμε κάθε φορά να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην οικονομία και στην ανάπτυξη των συμφωνιών μας πριν τις ε, αναθεωρήσουμε ή πριν τις ανανεώσουμε. Υπάρχουν ρήτρε που αφορούν τη διαφάνεια, που αφορούν τον διαχωρισμό της χρηματοδότησης ε, αυτής ε, της αναπτυξιακής σε σχέση με τη συμφωνία και όσον αφορά την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των εθνικών κοινοβουλίων πρέπει να ξέρετε ότι τις περισσότερες φορές τα εθνικά κοινοβούλια συμμετέχουν καθότι κυρώνουν. Υπάρχουν ε, μέσα μαζικής ενημέρωσης στις χώρες αυτές. Υπάρχει τύπος, ελευθερία έκφρασης και πολλές φορές διαβάζουμε με πολύ αρνητικό ή θετικό τρόπο ε, την περιγραφή της πολιτικής μας. Υπάρχει λοιπόν πραγματική συνειδητοποίηση και συζήτηση όσον αφορά τις αρνητικές ή ε, θετικές επιπτώσεις αυτών των συμφωνιών. Σας ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε, λέει ο να δώσω το λόγο και στον ε, συνάδελφό μου από την ε, ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να πω και εγώ δύο λόγια. Όπως υπόθηκε, η έκθεση αυτή μας βοήθησε να εντοπίσουμε κάποιες αδυναμίες ε, και ασυνέπειες στην κοινωνική πολιτική σε ό,τι αφορά την αλληλεία είναι πολύ σημαντικά. Τα συμμετόπαια εντοπίστηκαν, όπως γνωρίζουμε όλοι, η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αλία είναι ένα εργαλείο για την καταπολέμηση της ε, έλλειψης ασφάλειας στον τομέα των ε, τροφίμων. Εμείς ε, ως ΓΑΜΑ θα δώσουμε μεγάλη προσοχή στο θέμα αυτό στο πλαίσιο του προγραμματισμού μας και σε ορισμένες χώρες Θέλουμε να συμπεριλάβουμε την ασφάλεια των τροφίμων και την αλληλεία στους τομείς προτεραιότητας για τη συνεργασία. Και βέβαια θα, θα εργαστούμε μαζί και με τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΜΑΡΕ προκειμένου να Προκειμένου λοιπόν να καθορίσουμε τις ε, πολιτικές και στο πλαίσιο των αλληλευτικών συμφωνιών αλλά και του καθορισμού των προτεραιοτήτων στο πεδίο της συνεργασίας μας με αναπτυσσόμενες χώρες. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι στο πλαίσιο του προγραμματισμού για το 2014 στο 2020 η Γενική μας Διεύθυνση προσπαθεί να δώσει έμφαση στην ασφάλεια των τροφίμων και στο σκέλος Αλία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στον κύριο Φερέιρα, λέει ο πρώτος, για να ολοκληρώσουμε με τη συζήτηση του αυτού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους για την ε, συμβολή στη συζήτηση και τις προτάσεις ε, που ακούστηκαν. Πιστεύω ότι κάποιες από αυτές μπορούν πραγματικά να επιλουτίσουν αυτή τη γνωμοδότηση. Ξέρετε, να σας θυμίζω ότι 1500 χαρακτήρες ε, είναι ο περιορισμός ε, για την σύνταξη μιας ονομοδότησης. Άρα ε, δεν μπορούσα να επεκταθώ περαιτέρω, αλλά πιστεύω ότι θα εμπλουτίσει το κείμενό μου με τις τροπολογίες σας. Σε ό,τι αφορά τον απολογισμό, ε, σε ό,τι αφορά θετικές και αρνητικές συνέπειες. Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές οι συμφωνίες συνεργασίες αφορούν ένα πολύ, πολύ μικρό κομμάτι της αλληλευτικής δραστηριότητας αυτών των χωρών. Συμφωνώ που να γίνει ένα απολογισμό και να λαμβάνουμε πώ είναι και τι θετικέ και τι αρνητικέ συνέπειε. Αλλά αν θέλουμε να αποτιμήσουμε τι συμφωνίε και να τι βελτιώσουμε στο μέλλον, πρέπει να ξεκινήσουμε από μία διαπίστωση ότι αποτελέσματα μπορεί να έχουν από το επιθυμητό. Και επισημάνω κι εγώ κάτι θετικό, όπως αυτά που είπατε και εσείς. Ε, ε, εγώ δεν έχω καμία διαφορά υπάρχουν θετικά στοιχεία, αλλά επαναλαμβάνω που έχουν από τον ε, τελικό στόχο, ιδίω σε ό,τι αφορά τον ελληνικό κλάδο για αυτές τις τρίτες χώρες. Βεβαίω, δεν μπορεί να αναπτυχθεί ένα τέτοιο οικονομικό κλάδο μια μέρα στην άλλη, αλλά να σα υπενθυμίσω ότι χώρε όπω η Μαυριτανία, που ουσιαστικά αφο, για αυτή τη χώρα αφορά την πλέον σημαντική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει συμφωνία. Δεν έχει νέο συμφωνία το 2004 και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθο, εδώ και δύο δεκαετίε αυτή η συμφωνία με την Βρετανία προβλέπει και μία α, διάσταση συνεργασία σε αυτό το τομέα. Δεν θα έπρεπε λοιπόν επιτόπια να πάει η Κομισιόν στη Μαρτανία για να δει ποια είναι τα αποτελέσματα μιας τέτοιας συμφωνίας ε, εδώ και δύο δεκατιών. Ε, πώς να μην το πει κανεί για να διαπιστώσει τελικά ότι τα τελικά αποτελέσματα ε, απέχουν πολύ από τις αρχικές επιθυμίες. Και εδώ μιλάμε για πολιτική δύο δεκατιών και δεν μιλάμε για μεγάλη βιομηχανία, για ένα λιμάνι. Ένα λιμάνι Ούτε μιλάμε ε, για μια χώρα με τεράστιε ακτογραμμέ. Η Μαυρτανία έχει μόνο ένα λιμάνι στο βορρά και 700 χιλιόμετρα ακτών και στις 20, στα 20 έτη στην αυτή χώρα δεν καταφέρουμε να έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα. Θέλω να πω ότι ενώ ναι, μένω συνολικά. Και εγώ φυσικά δεν θέλω να παραβλέψω τις θετικές συνέπειες, το θετικό αντίκτυπο αυτών των συμφωνιών, αλλά στην πράξη τώρα στη συνεργασία πόρο απέχει από ε, το ποθητό. Αυτές οι συμφωνίες κατά κύριο λόγο γίνονται με τρίτες ανάπτυξη χώρα. Κάποιες φορές έχουμε και συμφωνίες με τις ε, ελάχιστε αναπτυγμένες χώρες. Χώρες ε, που, αν θέλετε, οι πόροι, η οικονομική βοήθεια που προβλέπουν αυτές ε, οι συμφωνίες αποτελούν πολύ σημαντική οικονομική στήριξη για τον προπολογισμό των χώρων αυτών. Είναι πολύ σημαντικές συμφωνίες λοιπόν για αυτές τις χώρες και δεν πρέπει να το παραγνωρίσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Φερέιρα. Ολοκληρώνει τη συζήτηση επί του σημείου αυτού και περνάμε στο επόμενο σημείο της διάταξης. Τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου που προβλέπει μακροπρόθεσμο σχέδιο για τα αποθέματα γάδου και τις αλλιευτικές δραστηριότητες που μεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά. Ο πρόεδρο, συγγνώμη, αλλά ξέχασα να σα πω κάτι σε σχέση με το προηγούμενο σημείο. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών λήγει στι 16 Ιουλίου και ώρα 12 το μεσημέρι. 16 Ιουλίου. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών για την έκθεση Φερέιρα. Ay, perdón. Es el informe de la señora Dodds y vamos a tener... Λοιπόν, πρώτη ανταλλαγή απόψε είναι εκθέσεως Dodds, σημείο 18. Δίνω το λόγο στην κυρία Dodds. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που βάλατε στη μεσή διάταξη ε, νωρίτερα την ανταλλαγή απόψεων για αυτό το θέμα. Ήταν ε, μία περίοδος που είναι ιδιαίτερα πολύ άσχολη από τότε που πρώτο συζητήσαμε το θέμα αυτό στην Επιτροπή στον προηγούμενο μήνα και υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία διακυβεύονται. Θα ήθελα λοιπόν να τα σκιαγραφίσω με πολύ απλό τρόπο και εν συντομία. Ο κανονισμός ε, του Συμβουλίου 1342 θεσπίστηκε το 2008 πρόλης Λισαβόνας Επομένως είναι σαφές ότι υπάρχουν αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στον κανονισμό αυτό, τόσο ώστε να προσαρμοστεί με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτή είναι μία από τις ευθυγραμμίσεις που θα πρέπει να συμφωνηθούν μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, μεταξύ άλλων. Ωστόσο, φαίνεται, στο γενικό πλαίσιο των ευθυγραμμίσεων αυτών, ότι ε, δεν είναι πάρα πολύ σαφή η διοργανική συμφωνία, το αντίθετο μάλιστα. Και ακόμη και αν είχε ολοκληρωθεί σήμερα στην Επιτροπή μας αυτή η ευθυγράμμιση, θα κολούσε αν θέλετε μετά ε, σε μια μεγάλη ουρά άλλων θεμάτων ε, στο πλαίσιο της διελκυστίδας που υπάρχει για το πώς θα εντάξουμε στους κανονισμούς της διαδικασίας της συνθήκες της Λισαβόνας. Από ό,τι γνωρίζω, σημειώθηκε μικρή πρόοδος, πρόοδος πάντως, στο θέμα αυτό επιδανικής προεδρίας. Γνωρίζω ότι οι συνάδελφοι της Επιτροπής αυτής έχουν και αυτοί εκθέσεις ε, που περιμένουν στην ουρά, στην μακριά, μεγάλη αυτή ουρά. Και φυσικά ξέρω ότι πολλοί αγωνιούν για να υπάρξει πρόοδος σε αυτό το θέμα και σίγουρα θα το θέσω και εγώ ως προτεραιότητα σήμερα στον ε, Κύπριο Υπουργό. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να σημειώσουμε πρόοδο στο σκέλος αυτό της έκθεσης, αλλιώς δεν πρόκειται να προχωρήσουμε, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε σήμερα να μας ενημερώσει σχετικά με το πώς οι ίδιοι ε, αντιλαμβάνονται την πρόοδο, αν έχει σημειωθεί πρόοδος, και επί της Κυπριακής Προεδρίας. Πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είχαμε λοιπόν ένα πρόβλημα με την ευθυγράμμιση. Δεν είναι κάτι το οποίο η Επιτροπή μας ε, πρέπει να το δεχθεί. Πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο. Πρέπει να προχωρήσουμε μαζί και με τους άλλους παράγοντες της όλης διαδικασίας. Και αυτό θέλω να το θέσω όλους ε, να είναι πολύ ξεκάθαρο. Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτή την ευθυγράμμιση, υπάρχουν κάποια πράγματα που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό που θέλουμε να δούμε είναι η νομοθετική διαδικασία που είναι σημαντική να ενσωματωθεί στην όλη διαδικασία. Και τα δύο σκέλη της νομοθετικής αρχής, Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, να έχουν ε, τη θέση τους σε αυτή τη διαδικασία ευθυγράμμιση. Εγώ βλέπω και κάποιο χώρο για τις ε, κατεξουσιοδότηση Είναι κάτι που το ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σχετικό της έγγραφο. Εγώ θεωρώ ότι οι κατεξουσιοδότηση πράξης μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα, σε αυτό το σχέδιο και πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι πλέον υπάρχει μια μετατόπιση αντί των ε, ξεχωριστών σχεδίων και προγραμμάτων να προχωρήσουμε, θα ήθελα εγώ τουλάχιστον, ε, σε κάποια προγράμματα που να περιλαμβάνουν πολλά είδη, πολλαπλά είδη και έτσι θα έχουμε μια συνολική εικόνα της κατάστασης. Είναι σημαντικό λοιπόν το πώς θα αναπτυχθεί αυτό το σχέδιο τα επόμενα χρόνια. Στο άρθρο 10 Τη πρόταση ε, περιθωράμισης βλέπουμε να λέει η Κομισιόν ότι κατά εξουσιοδότης πράξη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προσαρμογές ε, σε επίπεδο βιολογικής αναφορά ε, σε ποσοστά θνησιμότητας ψαριών, δείκτες κτλ. Είναι σημαντικό, θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε σημαντικά τα σχέδια και η όλη νομοθετική διαδικασία δεν μπορεί να το κάνει αυτό από μόνη της. Θέλω λοιπόν να ξεκαθαρίσω ότι εγώ βλέπω να έχουν θέση η καταξιοδότηση πράξης και είναι σημαντικό, σημαντική η θέση τους. Η Επιτροπή μας όμως προτού δώσει αυτή την δυνατότητα για τη κατεξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να καταστήσει απόλυτα σαφές τι θέλει να περιλαμβάνουν αυτές τις πράξεις, μέχρι πού μπορούν να πηγαίνουν, ποιο θα είναι το πεδίο εφαρμογή του. Για παράδειγμα, θα με ανησυχούσε αν στην πρόταση αυτή ε, η της πράξη συνέχιζαν να εξετάζουν τα αλληλευτική προσπάθεια. Πρέπει να είναι πολύ σαφή λοιπόν τα πράγματα, τα όρια των της πράξεων ε, και το πεδίο εφαρμογή τους. Εδώ ε, σταματώ πάνω σε αυτό και θα ήθελα να ακούσω και τις απόψεις των συναδέλφων για αυτό το θέμα. Έτσι θα προχωρήσουμε σε αδρές γραμμές και βέβαια θα δούμε και στην επόμενη σύνοδο, ε, στην επόμενη συνδρίαση ε, και το σχέδιο έκθεση που θα σας παρουσιάσω. Υπάρχει όμως και ένα τρίτο θέμα, σημαντικό, για τη συζήτηση που θα έχουμε τις επόμενους, ε, που θα έχουμε τις επόμενες, τα επόμενα λεπτά. Υπάρχει αυτή η καθυστέρηση οργανική, όπως είπα, και αυτό ο αγώνας εξουσίας. Εγώ δεν ξέρω να υπάρχει τεράστιο. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε αυτή την ευθυγράμμιση και φαντάζομαι ότι συμφωνούν όλοι ότι οι περισσότεροι τουλάχιστον ότι πρέπει να τροποποιηθεί και μάλιστα κατεπηγόντω ο κανονισμό. Οι επιστήμονες και αυτοί συμφωνούν ότι κάποιες ε, τροπολογίες ε, είναι απαραίτητε για τον κανονισμό αυτό. Σε ό,τι αφορά ε, τη βιώσιμη αλία, την προστασία των αποθεμάτων και ελπίζω επίσης μπορεί να βοηθήσει αυτό και στο να είμαστε επιλεκτικοί σε ό,τι αφορά τα αληφτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται. Υπάρχουν λοιπόν τρόπο που θα μπορούσαμε να προωθήσουμε προς αυτό το στόχο. Και επειδή στην προηγούμενη παρουσίαση από την Κομισιόν αναφέρθηκε, θα ήθελα να μου πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι χρονοδιάγραμμα προτείνει για την κατάσταση αυτών των τροποποιήσεων. Στο γραφείο μου, μαζί με το προσωπικό μου, ε, είχαμε μια συνάντηση τον Ιούνιο και εκεί μου είπαν ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την ε, κατάθεση τροπολογιών για τον κανονισμό. Κανένας λοιπόν δεν μπορούσε να μου δώσει καμία ένδειξη για το πότε θα μπορούσαν να προταθούν τέτοιες τροποποίησεις. Το μόνο που πρέπει να γίνει ουσιαστικά να προχωρήσει αυτή η διαδικασία ευθυγάμισης, από τις ξέρετε, συμφωνούμε, αλλά δεν βλέπω να πηγαίνουμε πιο πέρα. Δεν μπορούμε εμείς να το θέσουμε σε ισχύ, να το ενεργοποιήσουμε. Και πραγματικά καταλαβαίνετε πόσο αναστατώθηκα όταν αργότερα που μου είχαν πει από την Επιτροπή Σφεξέλης ότι δεν υπάρχει προθεσμία για τροπολογίες, δεν υπήρχαν τροπολογίες και δεν υπήρχε ε, χρονοδιάγραμμα. Ξαφνικά, σε μια συνάντηση στο Δημβούργο των κλάδων και των επιστημόνων, συζητούνταν αυτές οι τροπολογίες για αυτόν τον ε, κανονισμό. Και τι έχω μαζί μου, τις τροπολογίες αυτές, για τους συναδέλφους. Θα σας τις διαβιβάσω κύριε Πρόεδρε, ώστε με τη διακριτική σας ευχέρεια να τις διανύμετε στους συναδέλφους. Πραγματικά ε, δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένη. Εμείς κάνουμε εδώ την δουλειά μας ολιστικά, όπως θα επιθυμούσαμε. Δεν έχουμε σαλαμοποιήσει τα πράγματα, ούτε τα έχουμε βάλει όλα βέβαια στο ίδιο τσουβάλι, αλλά είδαμε ότι τελικά έγινε μια συνάντηση του κλάδου στην, στο Εδιμβούργο με τους επιστήμονες και συζητήθηκαν τροπολογίες συγκεκριμένες εκεί. Θα σταματήσω εδώ. Νομίζω ότι η Επιτροπή, σας, ε, Επιτροπή μας πρέπει να ανησυχήσει ιδιαίτερα για την εξέλιξη αυτή. Οι τροπολογίες ε, φυσικά και έχουν δημοσιοποιηθεί, αλλά θα έπρεπε πρώτα να τις είχαν ε, λάβει οι συνομοθέτες και οι βουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου. Φαντάζομαι ότι είναι ένα θέμα που θα θέλει η Επιτροπή μας να το συζητήσει. Συνοπτικά λοιπόν, τρία σημεία βλέπω. Τρία στοιχεία σε αυτά που κάνουμε. Πρώτο, πρόκειται για μια διαδικασία. Αυτή ε, η διαδικασία σχετίζεται άμεσα με αυτή τη διελκυστίνδα που υπάρχει για το πώς θα γίνουν οι ευθυγραμμίσεις με την Λισαβόν. Δεύτερον, νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε με την νομοθετική διαδικασία και την ευθυγράμμιση. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Νομίζω ότι οι συνάλφοι εδώ μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με το πώς θα προχωρήσουμε. Και τρίτον, εν ώψη του ότι υπάρχουν ε, και έχουν δημοσιοποιηθεί τροπολογίες, πρέπει να δούμε πώς αυτό θα προχωρήσει και σε σχέση με τον κανονισμό. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη αν έχω μακρηγορήσει λίγο, αλλά είναι θέματα σημαντικά. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Τότς. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Λεπέν που ζήτησε το λόγο ή προτιμάτε να ακούσετε την ε, Κομισιόν πρώτα. Να δώσουμε πρώτα το λόγο στην Επιτροπή, στην κυρία Μοντέση. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την ε, κυρία Τότς για την ε, παρουσίαση της. Αν μου επιτρέπετε, να διευκρινίσω κάποια σημεία όπως ζήτησε η εισηγητρία. Είχαμε την ευκαιρία να σας εκθέσουμε την πρότασή μας στην τελευταία συνεδρία της Επιτροπής σας και να πούμε ότι αυτή η πρόταση είναι μία πρόταση που απορρέει από την διοργανική ε, συμφωνία, με στόχο δηλαδή την ευθυγράμμιση. Κάτι που κρίθηκε αναγκαίο και ήταν υποχρέωσή μας λοιπόν να προτείνουμε αυτή την ευθυγράμμιση. Βεβαίω απορρέουν ε, και κάποιε ερωτήσει σχετικά με το ποιο είναι υπεύθυνο γιατί και κατά πόσον ε, το κατάλληλο εργαλείο είναι πράξη καταξιοδότηση ή όχι. Είναι ένα θέμα που συζητείται και παρακολουθούμε βεβαίως και τέτοιες απόψεις. Η κυρία τότε είπε ε, μεταξύ άλλων ότι είναι αναγκαίο να γίνουν και παρακολουθουμε βεβαιως και δικέ αποψει η κυρια τοτε ειπε μεταξυ τροποποίησεις στο πρόγραμμα για τον γάδο. Όπως είχαμε την ευκαιρία να σας επενθυμίσουμε και στην τελευταία συνεδρίαση, ήδη έχει δρομολογηθεί μία δραστηριότητα στην ε, Σκόλπους Επιτροπής για να γίνουν σχετικές τροποποιήσεις. Άρα λοιπόν, εμάς δεν μας εκπλήσει ε, το γεγονός ότι λάβατε κάποια ενημέρωση για μία συνεδρίαση στο Εδιμβούργο. Ε, εκεί θα συνεδριάσει, μάλλον εκεί συνεδρίασε η Επιστημονική Επιτροπή στην οποία υποβάλαμε με πλέον διαφανή και δημόσιο τρόπο κάποια στοιχεία που ζητούμε την ε, επιστημονική τοποθέτηση της Επιστημονικής Επιτροπής για να τα λάβουμε υπόψη κατά τροποποίηση του σχεδίου αποκατάσταση του γάδου. Λοιπόν, μετά από κάποια αιτήματα, ερωτηματικά που είχαν συμπεριληφθεί στην ε, αξιολόγηση ε, για το πρόγραμμα κατάσταση του γάδου και με βάση και τις συζητήσει που έλαβαν χώρα στο Συμβούλιο τον περασμένο Δεκέμβριο, ήδη είχαμε ανακοινώσει, δημοσίω, δηλαδή, ότι επεξεργαζόμαστε μία προσπάθεια πρόταση, συγγνώμη, τροποποίηση του κανονισμού για το γάδο, ώστε να τον απλοποιήσουμε, ιδίως σε ό,τι αφορά τις ελευτικές προσπάθειες. Πρόκειται λοιπόν για μία δραστηριότητα που έχει δρομολογηθεί, είναι σε εξέλιξη, γίνεται με τον κλάδο, με τη βοήθεια της Επιστημονικής Επιτροπής και σε επίπεδο ε, ομάδων εμπειρογνωμών που ήδη έχουν συνδυάσει πολλές φορές και είμαστε σχεδόν στην τελική φάση. Η πρόταση κανονισμού είναι στη διαδικασία έγκρισης στα πλαίσια της Επιτροπής. Κύριε Δότ, δεν μπορώ να δεσμευθώ σε κάποιες ημερομηνίε. Ακολουθούμε τη, τους κανόνες που ισχύουν στις περιπτώσεις, αλλά σίγουρα είναι αυτό το χρόνο θα υποβληθεί υπόψη σας και βεβαίως θα είναι και πάλι χαρά μας να σας παρουσιάσουμε σε κάθε λεπτομέρεια τις προτάσεις τροποποίησης που θα ε, υποβάλουμε από εκεί πέρα λέω ότι δεν μπορώ να πω κάτι για ημερομηνίε, γιατί η διαδικασία λήψη αποφάσεων και έγκριση πρόταση είναι σε εξέλιξη. Πάντω, σύντομα, σύντομα θα έχετε αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Μοντέση. Κυρία Λέβεν. Ε, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Ντότ για την έκθεσή της. Συμφωνώ με την πρώτη εκτίμηση που κάνατε. Όντως, φτάνουμε σε κάτι το εντελώς παράλογο. Πρόκειται για μια ευθυγράμμιση διαχειριστικών σχεδίων, συνδιονάκτησης ε, διαφόρων ε, τομέων, ευθυγράμμιση με αυτά που προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας. Και εδώ, σαφώς και αν συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο, θα πρέπει να επιτευχθεί πάρα πολύ γρήγορα μια συμφωνία και ε, το χρειαζόμαστε. Δεν μπορούμε να έχουμε μακροχρόνια διαχειριστικά σχέδια για όλα αυτά τα αποθέματα. Συμφωνώ λοιπόν απολύτως μαζί σας ότι το θέμα υπήγει και ότι το θέμα των κατεξουσιοδότηση πράξεων είναι ανάγκη. Δεν μπορούμε δηλαδή μονίμως να ενεργοποιούμε τη διαδικασία της συναπόφασης για όλα τα θέματα. Αλλά βεβαίως με τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξεις αναθέτουμε τις αρμοδιότητες σε κάποιον άλλον. Δεν μπορούμε να εκφραστούμε σαν κοινοβούλιο. Και εδώ αρχίζω να ανησυχώ αν θέλετε. Γιατί όπως έχει σήμερα η κατάσταση, οι σχέσεις μας με το Συμβούλιο, θα πρέπει ναι με να ευθυγραμμιστεί, αλλά και να αλλάξει και να τροποποιηθεί ε, ένα μεγάλο τμήμα αυτών των σχεδίων. Και νομίζω ότι συμφωνείτε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, ανάγκη βελτίωσης. Δεν γνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες, αλλά ξέρω ότι σαφώς και υπάρχουν εδώ τροπολογίες οι οποίες θα πρέπει να υποστηριχθούν από μας. Σαν αρχή, αν θέλετε, είναι θέμα αρχής, ανησυχώ λίγο καθότι οι σχέσεις μας θα γίνουν ακόμα πιο περίπλοκες με το Συμβούλιο. Και για να φτάσουμε σε μια συμφωνία, ίσως δεν θα πρέπει σε αυτό τουλάχιστον το στάδιο να ε, προτείνουμε πολλά νέα στοιχεία. Ας περιμένουμε, αν θέλετε, να φτάσει μία πρόταση για ένα νέο διαχειριστικό σχέδιο στο Κοινοβούλιο και κατόπιν υποβάλλουμε τις τροπολογίες μας. Αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Οι σχέσεις μας με το Συμβούλιο. Γι' αυτό και εγώ θα πρότεινα να είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί ως προς τις ε, τροπολογίες αυτών των διαχειριστικών σχεδίων και θα αναφερθώ και στο θέμα των αλλιευμάτων στην Βαλτική, του γάτου στη Βαλτική. Προσωπικά λοιπόν θα παρέμενα σε αυτήν την ευθυγράμμιση και θα περίμενα ε, τη νέα πρόταση για να υποβάλουμε περισσότερες ε, τροπολογίες. Και αυτό ισχύει και για την Βαλτική και για τη Βόρεια Θάλασσα, για το Γάδο. Κάνατε και μία ερώτηση. Γιατί δεν σας ενημέρωσαν ενώ είστε η συγγήτια. Έχετε δίκιο. Βεβαίως και υπάρχει υποχρέωση να ενημερώνεται ο εισηγητής σε όλα τα στάδια της ε, διαδικασίας μέχρι να φτάσουμε στο νέο σχέδιο. Γιατί εμείς είμαστε οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των πολιτών και είναι αυτονόητο ότι πρέπει να ενημερωνόμαστε. Ευχαριστώ κύριε Ρόδους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ την κυρία Ντάτση για την πολύ ειλικρινή και ανοιχτή παρουσίασή της αυτά που μας ενημέρωσε. Ε, πραγματικά με κάνουν να ανησυχώ. Εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξη όπως η κυρία Λεβεν. Εδώ και τέσσερα χρόνια δεν έχει αποφασιστεί κανένα πολιετές σχέδιο. Και ε, μονίμως ακούμε ότι γι' αυτό φταίει το Κοινοβούλιο. Κοιτάξτε, εγώ πραγματικά εκπροσώπησα το κοινοβούλιο στο Βερολίνο όταν άκουσα τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου να λέει ότι όλα αυτά οφείλονται στη στάση του Κοινοβουλίου. Λοιπόν, κοιτάξτε, εμείς έχουμε εκφραστεί και θα ήθελα η κυρία Ντότς πραγματικά να μας ε, εκφράσει και γραπτός αυτά που μας είπε εδώ γιατί πραγματικά θεωρώ ότι εδώ πρέπει να ζητήσουμε συμβουλή από την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου για να δούμε επιτέλους τι δυνατότητες έχουμε έτσι ώστε να σταματήσει αυτό το παιχνίδι πλέον. Είναι πραγματικά τραγικό το ότι στην κοινή γνώμη το Συμβούλιο συνεχίζει να λέει ότι εμείς είμαστε υπέτειοι για αυτές τις αποτυχίες. Ε, φτάνει πια αυτό. Και δεν είναι δικαιολογημένα αυτά που ακούγονται. Γι' αυτό και νομίζω ότι πρέπει επιτέλους να αντιδράσουμε. Και γρήγορα. Ευχαριστώ. Κύριος Κάλαγκαρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ την κυρία Τότς. Ε, φαίνεται ότι έχει κάνει πολλή έρευνα για αυτό το θέμα, όπως συνηθίζει να κάνει. Να ένα ακόμη από αυτά τα προγράμματα αποκατάστασης είναι σημαντικά αυτά τα προγράμματα, ιδίω αυτό αφορά την αποκατάσταση του γάδου. Ε, ναι, αυτό είναι το σημείο εκκίνηση ε, που είχαμε πάντοτε, ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτά τα μακροχρόνια προγράμματα αποκατάστασης για να υπάρχει βιωσιμότητα. Χρειάζεται λοιπόν ένα τέτοιο πρόγραμμα. Ε, ευτυχώς έχουμε φύγει από την εποχή των ad hoc ε, προγραμμάτων και οικονομικός πώς μακροχρόνια προγράμματα μπορούν να λειτουργήσουν. Μας ε, απίθανε και το σχετικό ερώτημα στη χώρα μας σχετικά με το πώς λειτουργούν αυτά τα προγράμματα και προσπαθούμε να εξηγήσουμε ότι πραγματικά δεν μπορούμε να αποφασίσουμε σε τίσια μόνο βάση. Θα πρέπει να έχουμε μακροχρόνια, μακρόπνοα προγράμματα για να υπάρχει και ένας μακροχρόνιος σχεδιασμός. Και εγώ ήμουν θύμα. Ε, δεν θα αναφερθώ λεπτομερώς, όπως τόσε συνάδελφοι, κύριε Παπά, κύριο Στίβενσον και η κυρία Τότς. Ε, έχουμε υπάρξει θύματα της παραπληροφόρησης. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να το θέσουμε αυτό, πρόεδρε. Ε, να σας πω ότι... Ξέρετε, σε πρόσφατη συνάντηση που είχαμε την πρώτη του Κοινοβουλίου, με εξέπληξε και με την θέση του και τη βούλησή του, ο οποίος είπε ότι θα μιλήσει και με τον ε, Κύπριο Πρόεδρο, θα το θέμα ότι θα πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη επικοινωνία και πληροφόρηση και πιστεύω να αποσταλεί ένα σαφέ μήνυμα προ την Κυπριακή Προεδρία. Ανεξάρτητα από τα θέματα που θα απασχολήσουν την Κυπριακή Προεδρία, ιδίω για αυτό το θέμα, θα πρέπει να υπάρξει πρόοδο. Ε, θα πρέπει να επενέσουμε τη Δανική Προεδρία, τον τριμερή διάλογο που είχαμε και συμφωνούμε, πιστεύω, όλοι ότι αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το προωθήσουμε. Ε, είμαστε ρεαλιστέ. Πράξη κατοξιοδότηση είναι μια ρεαλιστική πρόταση. Δεν μπορούμε να κάνουμε μικροδιαχείριση σε αυτό το θέμα. Θα είμαστε λογικοί στι απαιτήσει μα. Και βεβαίω, εγώ μόνο για τη δική μου έκθεση μπορώ να μιλήσω. Αλλά έχω την αίσθηση ότι και η Κομισιόν έχει ένα άγχος να ε, υπάρξει πρόοδο. Πιστεύω, Πρόεδρε, ότι όταν θα γραφτεί η ιστορία εκεί θα γραφτεί κατά πόσον έχουμε επιτύχει πρόοδο το, το, το επόμενο διάστημα. Ξέρετε, σε λίγα χρόνια θα έχουμε μια νέα του Κοινοβουλίου, θα έχουμε νέους ανθρώπους και θα μας κρίνουν πολύ σύντομα ότι δεν έχουμε εμφανίσει το ύψος των περιστάσεων. Θα πρέπει λοιπόν να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να υπάρξει πρόοδος. Ξέρετε, κυρία Τότς αισθάνεται θλίψη για τον τρόπο τον οποίο γίνονται οι ότι ενημερώθηκε μεν εκ των υστέρων ε, για πράγματα τα οποία άλλοι γνώριζαν πολύ νωρίτερα. Να κατανοώ ότι δεν χρειάζεται να υπάρξει ειδική ενημέρωση για το Κοινοβούλιο για κάποια ζητήματα, αλλά είναι καλό τουλάχιστον η εισηγήτρια, ο εισηγητή για ένα θέμα να ενημερώνεται. Ιδάλω δεν χρειάζεται καν να έχουμε επικοινωνία με την Κομισιόν γραπτός έχουμε τις προτάσεις τροποποίησης, άρα ποιο το νόημα. Πρόεδρε, πιστεύω ότι είναι ένα θέμα που θα μπορούσαμε να το ζητούμε όλη τη μέρα σήμερα. Μας απασχολεί όλους μας. Ίσως σε μια μελλοντική συνεδρία συντονιστών. Ίσως θα ήταν σκόπιμο να βάλουμε αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Ώστε να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να ορίσουμε έναν οδικό χάρτη να κάνουμε κάποια μελλοντικά βήματα, ώστε να μπορούν και οι συγκριτές στο μέλλον να ξέρουν που βαδίζουν. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ντότς, για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους και σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Θα σας περιγράψω όπως βλέπω τη διαδικασία από εδώ και πέρα, σύντομα. Το πιο σημαντικό σημείο είναι ότι δεν μπορούμε να προοδεύσουμε ό,τι και να κάνουμε. Δεν μπορούμε να προοδεύσουμε. Γιατί υπάρχουν κάποια στοιχεία που είναι εκτός της δικής μας αρμοδιότητας. Παρ' όλα αυτά, η Επιτροπή μπορεί να εκφράσει με σαφήνεια τις θέσεις της. Ευχαρίστως θα σας τα δώσω και γραπτά όπως μου ζητήσατε, θα τα δώσω στον Πρόεδρο και εσείς ε, κύριε Πρόεδρε μπορείτε να ενημερώσετε και ενδεχομένως αν ε, πρέπει να ζητήσουμε νομική συμβουλή στην νομική υπηρεσία γιατί όχι. Όσον αφορά τώρα την ε, υποβολή νέων στοιχείων, εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό θα δυσκολέψει τα πράγματα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε σύντομα είναι να υπάρξει εφηγράμμιση ας πούμε ότι η διαδικασία πρώτα θα ξεκινήσει με την ευθυγράμμιση και κατόπιν θα υποβληθούν τροπολογίες. Το θέμα όμως είναι ότι αυτή η ευθυγράμμιση είναι μια συνεχής διαδικασία, δεν θα σταματήσει ποτέ και ενδεχομένως θα μπορούσαν να είχαν ενσωματωθεί οι τροπολογίες σε αυτήν τη διαδικασία. Αν κοιτάξει κανείς τα στοιχεία που μας παρέχει το Συμβούλιο το Συμβούλιο θεωρεί όντω ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο να υπάρξει συμφωνία και για τις τροποποιήσεις ταυτόχρονα με το νέο πρόγραμμα. Δεν ξέρω. Θα επανέλθουμε πάντως σίγουρα στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τόντ. Μια ερώτηση μόνο για αυτό το ζήτημα έχω και εγώ είναι θέμα που το γνωρίζετε όλοι πολύ καλά. Τα μηνύματα, πιστεύω, έχουν περάσει με πολύ σαφήνεια. Και ευτυχώς ε, μιλάμε για ομόφωνα μηνύματα ε, που παίρνουν από πλευρά μας ε, προς την Κομισιόν. Η Κομισιόν έχει να αντιμετωπίσει μία ομόφωνη θέση του Κοινοβουλίου ο πρόεδρος Σούλτς ε, παρενέβη, τοποθετήθηκε η Κυπριακή Προεδρία. Ήδη είχαμε μια πρώτη συνάντηση και εγώ με τον ε, Υπουργό είχα μια συνάντηση και σήμερα το απόγευμα έχουμε τη συνάντηση με τον Κύπριο Υπουργό. Το μήνυμα είναι σαφέ. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ανεκτούμε, σε καμία περίπτωση, το Συμβούλιο να καταλήξει να ε, ρίξει την ευθύνη στο Κοινοβούλιο. Και το άλλο το Κοινοβούλιο έχει τοποθετηθεί, έχει ολοκληρώσει την πρώτη ανάγνωση. Το Συμβούλιο πρέπει να αναλάβει δράση. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν ε, μπορεί να στρουθοκαμιλίζει το, το, το, το Συμβούλιο. Α αποφασίσουν, α είναι θαραλέοι, α πούνε ναι ή όχι. Για να καταλήξουμε κάπου. Και αν ε, κρυθεί αναγκαίο, θα πάει το θέμα στο 10. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να φανεί ότι φταίει το κοινοβούλιο, το κοινοβούλιο που έχει κάνει τη δουλειά του, αυτό που το αναλογεί, και είναι κάτι που το έχουμε επισημάνει με κάθε σαφήνεια. Και έτσι κλείνουμε για αυτό το σημείο. Απλά θέλω να σας υπενθυμίσω κάτι άλλο. Μου είπαν σε ό,τι αφορά την γνωμοδότηση Φερέιρα, βάλαμε ως προθεσμή υποβολή τροπολογιών 16 του μηνός. Μου ζήτησαν να παρατείνουμε την προθεσμία στις 18. Άρα λοιπόν έως τις 18 ε, του μηνός το μεσημέρι υποβολή τροπολογιών για την γνωμοδότηση Φερέρα και το ίδιο του ε, θα σταματήσουμε τώρα και θα επιστρέψουμε στις 3 ακριβώς. Παρακαλώ να είσαστε ακριβείς γιατί έχουμε την, ε, πρέπει να υποδεχτούμε τον Κύπριο Υπουργό και με τον οποίο θα συζητήσουμε πολλά θέματα. Ευχαριστώ όλους θερμά. Θα ξαναπούμε στις 3.